Ως προς τη σειρά των εκθέσεων, η Άλντε ζητά η απόσπαση εργαζομένων να, να τεθεί σε ψηφοφορία στο τέλος, γιατί ένας από τους αναπληρωτές θα φτάσει καθυστερημένος. Ξεκινάμε λοιπόν με την έκθεση του κύριου Χρυσόγονου για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε. 21. I ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Είστε υπέρ, μάλιστα. Εγκρίνεται με μεγάλη διαφορά. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7, υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Είστε κατά μάλιστα. Είστε κατά. Άρα απορρίφθηκε. Γιατί έχουμε ισοπαλία. 11 όλα. Τώρα ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης ηλεκτρονικά παρακαλώ. Yes, uh, clearly adopted εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον κύριο Χρυσόγωνο. Και τώρα, σχέδιο έκθεσης του κυρίου Λεμπρετών Τεστ αναλογικότητας. Αξιολόγηση της αναλογικότητας. Η στολή έτοιμη. Τροπολογία 13. Υπέρ. 30. Κατά. Αποχές. Δεν. Δύο ακόμα. εγκρίνεται. Οπότε πάμε στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Ακόμα λείπει ένας. Να κλείσουμε την ψηφοφορία. Δεν εγκρίθηκε η έκθεση. Και τώρα η έκθεση της κυρίας Μπούτελαντ τροποποίηση τις οδηγίες 2004 37 για την, απόσπαση, για την προστασία μάλλον των εργαζομένων. Ενιαία ψηφοφορία. Γκούτελαντ. Νομική βάση. Παρακαλώ δύο ακόμα για να κλείσει η ψηφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Γκούτελαντ. Και τώρα ψηφίζουμε για την απόσπαση εργαζομένων. Εισηγητής ο κύριος Καβαντά. Τροπολογία 10 υπέρ κατά. Μπορούμε να κάνουμε έλεγχο. Ένας ακόμα πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θέλετε να ελέγξετε τροπολογία 8 Πέρας προφορίας εγκρίνεται υπέρ 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 10 υπέρ Ναι, είναι δύο-τρει σελίδε παρακάτω. Δέκα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114. Υπέρ. Α, είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά, αποχές, να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε. Παραδέχομαι ότι βλέπω λίγα χέρια να σηκώνονται. εγκρίθηκε 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ να κάνουμε έλεγχο για την 118 απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. Απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ 19 υπέρ, κατά. Να κάνουμε έλεγχο. Εγκρίνεται 20 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά μου να αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά να ελέγξουμε. Δύο ακόμα χρειαζόμαστε, πέρα στις ψηφοφορίες, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά να κάνουμε έλεγχο Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 και 60 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 και 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ Κατά. Έλεγχος για την 64. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Άρχεται. Λείπουν λοιπόν, ένα δύο ακόμα. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Συγχωρητήρια στον κύριο Καβαντά. Ωραία. Αυτό το ψηφίσαμε. Αυτές ήταν οι ψηφοφορίες.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 με το 27, 28 και 29 έλεγχος κατεξιοδότηση πράξεων και εκτελεστικών μέτρων όπου απλά σημειώνουμε Mr. you to, take the floor? Κύριε Τζαμπάσκι, θέλετε το λόγο? Okay. Now we take the joint items 12 uh, and... Λοιπόν, τώρα παίρνουμε τα σημεία 12 και 13 ανταλλαγή απόψεων και τον λόγο έχει ο κύριος Σάιερ ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχουμε πάλι μια νέα πρόταση για ευθυγράμμιση της νομοθεσίας με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Με συγχωρείτε κύριε Σάρη, λέει ο πρόεδρος. Ησυχία. Λοιπόν, μια που δεν είναι η πρώτη φορά που τα συζητάμε, μπορώ να είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω όπως ε, και την προηγούμενη φορά που με είχαν καλέσει στην διάσκεψη των Πρόεδρων ε, για το θέμα αυτό, πως 10 χρόνια μετά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας εξακολουθούμε να έχουμε αυτό το διορθωτικό πρόβλημα το οποίο σημαίνει ότι βασικά δημιουργείται εδώ μια κατάσταση στην οποία δύο ε, ισότιμα μέρη, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, δεν έχουν ε, ε, ξεκαθαρίσει τις αρμοδιότητες τους σύμφωνα με τη συνθήκη και ταυτόχρονα επικρατεί διχογνωμία. Και, και, όχι διχογνωμία, αλλά διαφέρουν και τα συμφέροντα γιατί το Κοινοβούλιο στις περισσότερες περιπτώσεις ενδιαφέρεται πάρα πολύ ειδικά μετά την ενημέρωση για τις πράξεις κατεξοδότηση που έχει αυξηθεί κατά πολύ την τελευταία δεκαετία. Το Κοινοβούλιο θέλει να γνωρίζει το τι συμβαίνει με την νομοθεσία που εγκρίνει και το τι θα συμβεί με αυτά τα ζητήματα. Ε, άρα δημιουργείται μια στασιμότητα Κάτι το οποίο σημαίνει ότι Συμβούλιο και Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνήσουν. Ε, αυτό το που κάνουμε τώρα είναι κάτι το διαφορετικό, αλλά έχουμε μία έκθεση και η δικιά μου έκθεση πριν από πολλά χρόνια, όπου είχαμε πει ξεκάθαρα και ποια είναι η διάκριση μεταξύ πράξεων κατεξοδότηση και κατεφαρμογή επί τη βάση αυτής της αρχής ε, για εμάς δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το ζήτημα είναι όταν πρέπει να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο, το οποίο σε περισσότερες περιπτώσεις ε, ε, θέλει να το αφήσει σε πράξεις κατ' εφαρμογή, γιατί τότε μόνο αυτοί μπορούν να ελέγχουν το τι συμβαίνει. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι θα έλεγα μια πρόβα, μια νέα φάση των όσων είχαμε πριν από λίγα χρόνια. Είχαμε τρία όμνιμπους, δεν θυμάμαι. Τι έγινε πριν από τόσα χρόνια. Η Κομισιόν είναι κάπως ουδέτερη εδώ, αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα από τα... στα περισσότερα σημεία τα κριτήρια διάκρισης είναι παρόμοια με τα δικά μας και εδώ συμφωνούμε, αλλά υπήρχε μια πρόταση τριών όμνιμπους που έπεσε θύμα της απορρίθμισης. Ε, κάτι το οποίο εγώ θεωρώ λάθος, το είχα πει τότε, αλλά ταυτόχρονα δεν ε, ήταν απλά κάτι το οποίο διέγραψαν, αλλά ήταν ε, γύρω στην εποχή που δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο. Ξεκινούσαμε διαπραγματεύσεις ε, και δεν ε, τα καταφέραμε τελικά. Έχει περάσει πολύς ε, χρόνος, οπότε τώρα μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε. Εν τω μεταξύ όμως η υπόθεση αυτή συνεχίζεται στο Κοινοβουλίο, οι επιτροπές, ειδικά στον τομέα της νέας νομοθεσίας, εφαρμόζουν αυτά τα κριτήρια και βεβαίως ε, τρώμε πολύ χρόνο εκεί πέρα και τώρα έχουμε τις ε, διαπραγματεύσεις. Δεν ήταν εύκολο. Αναβλήθηκε η συνεδρία στην προηγούμενη εβδομάδα. Και τώρα υπάρχει κάποια ελπίδα. Αυτά μπορούν να γίνουν μαζί γιατί τι κάνουμε εμείς. Με βάση τη νέα πρόταση της ε, Κομισιόν έχουμε δύο πακέτα ε, που ευθυγραμμίζονται. Δηλαδή το ένα είναι βασικά νομικές αρμοδιότητες, ξεκάθαρα της ε, Γιούρη. Το άλλο είναι αρμοδιότητες άλλων επιτροπών στο Omnibus, οπότε υπάρχουν πολλοί κανόνες και αυτό βεβαίως το αναφέρω και στο εγγραφό μου. Ε, προτείνω δηλαδή να ακολουθήσουμε αυτό το οποίο είχαμε κάνει πριν από πέντε χρόνια, την ίδια προσέγγιση. Δηλαδή, εφόσον είναι ξεκάθαρο ήδη πως η Επιτροπή Γιούρη είναι η αρμόδια για την ευθυγράμμιση και ο λόγος ε, είναι σαφής ότι χρειάζεται μία ενιαία προσέγγιση ε, από πλευράς Κοινοβουλίου γιατί το Κοινοβούλιο δρά με βάση κάποια κριτήρια. Όμως και εγώ βλέπω ότι το Συμβούλιο δεν έχει κάποιες αρχές εδώ πέρα που ακολουθεί, απλά θέλουν τα πάντα. Τα πάντα να είναι πράξεις ε, κατά εφαρμογή. Εμείς ε, θέλουμε να διατηρήσουμε κάποια νομοθετική αρμοδιότητα. Συχνά οι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν τη νομική πτυχή και είναι η Επιτροπή μας αυτή η οποία προσπαθεί ε, να δημιουργήσει κάποια συνέπεια. Ναι, ολοκληρώνω. Και έτσι ε, η, η θέση μας ισχυροποιείται. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, αν είμαστε ενωμένοι, ακόμα και αν σε κάποιους κλάδους χάνουμε κάποιες τεχνικές δυνατότητες, αν είμαστε ενωμένοι, προσπαθούμε να έχουμε μια ενιαία θέση. Το συμπέρασμά μου είναι ότι η πρότασή μου εδώ ε, είναι να ακολουθήσουμε τη γραμμή που είχαμε και προσπαθούμε ακριβώς ε, να ενσωματώσουμε και τις γνωμοδοτήσεις ε, των επιτροπών που δεν έχουν κάποιο ειδικό καθώς. Λοιπόν, μας εμπιστεύονται καμιά φορά και με το τίμημα του να είμαστε υπερβολικά άκαμπτοι, αλλά θα ήθελα να πω πως ε, το μήνυμα θα περάσει και θα ήθελα να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία γιατί έχει αργήσει. Αλλά 10 χρόνια, έχουμε ήδη 10 χρόνια εμπειρίας. Εγώ θα ήθελα να μην έχουμε σε κάθε νομοθέτημα της ε, πράξης ε, κατεξουσιοδότηση και καταφαρμογή. και τους, τους επιτρέπουμε ακόμα και στην περίπτωση των πράξεων ε, κατά εξουσιοδότηση να κάνουμε την χειρονομία της καλής θέλησης. Αλλά στα γενικά κριτήρια περιέργως ακολούθησαν αυτήν την γραμμή και ελπίζω να το συνεχίσουν και τώρα. Ελπίζω να ολοκληρώσουμε πριν το τέλος του έτους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μπούντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Σάγερ για την παρουσίαση. Είμαι εισηγητής στην Επιτροπή Γεωργίας για τη γνωμοδότηση. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η προσέγγιση. Εγώ πρότεινα τροποποίηση των διοκανονισμών στην Επιτροπή Γεωργίας και πιστεύω πως όλες οι επιτροπές θα πρέπει να ασχολούνται μόνο με θέματα που άπτονται της εντολής τους. Πιστεύω ότι πρέπει να παρέμβουμε. Όμως πώς. Μέσω κατεξιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεων. Εγώ λέω μέσω κατεξιοδότηση πράξεων. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, εμείς έχουμε και την εμπειρία και τη γνώση για να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Δεν θα αμφισβητήσω την ε, ικανότητα της Κομισιόν να προβαίνει σε διευκρινήσει, αλλά θα ήθελα να ακούσω και την άποψη των υπόλοιπων συναδέλφων. Θέλει μήπως ο εκπρόσωπος της Κομισιόν και ο Κλάους να κάνει ένα σύντομο σχόλιο και βάζω δύο θαυμαστικά στη λέξη σύντομο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι είμαστε στη διάθεσή σας από οποιαδήποτε μορφή, είτε εδώ στην Επιτροπή σας είτε εκτός. Όπως είπε σωστά ο κύριος Σάγερ, αυτή είναι η δεύτερη απόπειρα να υπάρξει ευθυγράμμιση. Η πρώτη απόπειρα απέφυγε στο Συμβούλιο και είχαμε αποσύρει τότε την πρόταση γιατί δεν υπήρξε καμία κίνηση έκτοτε. Αυτό που θέλω να σημειώσετε είναι ότι τη φορά αυτή η πρόταση έχει μια σημαντική διαφορά. Έχουμε επιλέξει μια διαφορετική τεχνική. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε όλες τις εντολές μία προς μία και βλέπουμε και όλες τις νομικές ε, βασικές ε, πράξεις ξεχωριστά. Μιλάμε για 168 και νομίζω ότι υπάρχουν και 500 ε, εντολές, empowerments ε, ξεχωριστές. Άρα έχουμε ακολουθήσει πλέον την προσέγγιση ότι θα λάβουμε απόφαση για κάθε μία χωριστά. Αυτό που είναι σημαντικό για την Κομισιόν είναι αυτό που λέει η Διοργανική Συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία, την περσινή. Εκεί, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Κοινοβουλίου, λέμε ότι η ανάγκη ευθυγράμμιση ε, στο νομικό πλαίσιο που εισάγει η συνθήκη τη Λισαβόνα κτλ. Και τι είναι αυτό που εισάγει η συνθήκη τη Λισαβόνα, είναι ακριβώ αυτό το νέο πλαίσιο για εντολέ ε, που έχουν να κάνουν με δύο είδου ε, πράξεων. Έχουμε τις καθεξουσιοδότηση και τι εκτελεστικές πράξεις. Η επιλογή που έχει γίνει, που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή τη, είναι άκρο τεχνική ευθυγράμμιση Αμυγό τεχνική ευθυγράμμιση. Δεν αξιολογήσαμε καμία πρόταση εκχώρηση των empowerment, ε, ήταν πρόκειται να ε, γίνει, να μην γίνει κάποια εκτίμηση. Απλά περιοριστήκαμε στην τεχνική ευθυγράμμιση σε ό,τι αφορά είτε τις ε, κατεξοδότητες πράξεις εξεταλιστικές. Και Στι περισσότερε περιπτώσει, επειδή υπάρχει παρόν νομικό χαρακτήρα, επρόκειτο για κατ' κατεξοδότηση πράξη. Αυτά είχα να πω και προσβλέπω στη περαιτέρω συζήτηση και συνεργασία. Μάλιστα. Έχουμε πρόβλημα χρόνου. Γιατί... δεν καταφέραμε να δούμε τα δύο ζητήματα που είναι από χθε εξ και ρωτώ τους κυρίους ε, Ντελαβό και Τζαμπάσκη αν θέλετε να τα κάνουμε γρήγορα ή να τα αναβάλουμε. Η κυρία Ντελαβό ε, δεν έχει πρόβλημα με την αναβολή ούτε και ο κύριος Τζαμπάσκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε εγκαίρως ε, την ακροασή μας για την πρόταση περί αφαιρεγγιότητας και καλωσορίζω τους διακεκριμένους ε, προσκεκλημένους μας και χωρίς περαιτέρω εισαγωγή θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην κυρία Λετήσια Γκάγιο από την Τράπεζα BBVA της Ισπανίας, ε, επικεφαλής ε, του τμήματος κινδύνου και της νομικής υπηρεσίας που θα αναπτύξει το θέμα από τη σκοπιά των τραπεζών. Έχετε γύρω στα 10 λεπτά. So many thanks, Mr. Chairman. Ah, guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist wirklich ein Vergnügen, hier heute mit Ihnen zu sitzen. Σας ευχαριστώ. Είναι ευχαρίστηση και τιμή που είμαι εδώ πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ακρόαση και σας παρακαλώ να δείτε λίγο την παρουσίαση μπροστά ή πίσω σας, δεν ξέρω να κάνω μια εισαγωγή στην ε, BBVA. Βλέπετε, είμαστε μια μεγάλη ισπανική και ευρωπαϊκή τράπεζα. Έχουμε ε, δραστηριότητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα λέγαμε ότι είμαστε μια παγκόσμια τράπεζα. Και δεν είναι ρεαλιστικό βεβαίως να προσπαθήσουμε να δούμε ένα τέτοιο ζήτημα ε, σε 10 λεπτά μόνο. Θα ήθελα λοιπόν να εστιάσω σε κάποιες πτυχές του ζητήματος ε, που θεωρώ σημαντικές ε, από την ε, σκοπιά την δικιά μας αλλά και των πελατών μας που είμαι σίγουροι ότι θα επαναλάβουν και οι συνάδελφοι. Θα γνωρίζετε φαντάζομαι τις συστάσεις του Μαρτίου 2014 και της περσινής δημόσιας διαβούλευσης. Η Ισπανία όπως ξέρετε έχει εγκρίνει αυτήν την ε, σύσταση και μπορούμε έτσι να συμμετέχουμε κι εμείς στην ε, προτινόμενη αυτή ε, Ευρωπαϊκή Ένωση των Χρηματαγορών. Το υψηλό επίπεδο εφαρμογής της σύστασης μετά από μια δραματική αύξηση των χρεοκοπιών μας έχει οδηγήσει σε μια πάρα πολύ μεγάλη εστίαση σε αυτό το θέμα μετά από έναν μεγάλο αριθμό όπως είπαμε τέτοιων διαδικασιών γι' αυτό συμμετείχαν πάρα πολύ ενεργά στην διαβούλευση της ε, Κομισιόν Θα ήθελα λοιπόν να μάθω για αυτό το θα ήθελαμε να πούμε πως είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικέ οι προτάσει της Κομισιόν. Συγκεκριμένα κάποια πράγματα τα οποία έχουν ήδη δοκιμαστεί στο ισπανικό σύστημα και μοντέλο. Παραδείγματο χάρη, έχουμε πολλές και επικοινόμορφες διαδικασίε και ε, δικαστικές και εξοδικαστικές ε, ή με την εποπτεία του δικαστηρίου και θεωρούμε ότι έτσι μπορούν οι οφειλέτε να επιλέξουν μια διαδικασία που του ε, βολεύει περισσότερο και ανταποκρίνεται στο μέγεθος και την περιπλοκότητά τους. Όσον αφορά τώρα τη ε, διαδικασία αναδιάρθρωσης, ε, πέρα από την δικαστική τέτοια, έχουμε και μια δικαστική τέτοια διαδικασία που είναι πολύ επιτυχής όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το κλειδί της επιτυχίας είναι ότι πρόκειται για μια ευέλικτη διαδικασία, δεν εμπλέκονται τα δικαστήρια, δεν υπάρχουν καθυστερήσει και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Όσον αφορά τώρα τις ε, διαδικασίες εντός του δικαστηρίου θεωρούν ότι θα πρέπει να, γίνουν, να γίνει διάκριση μεταξύ δύο ειδών πιστώσεων, τις ασφαλισμένες και μη. Ε, Μπορεί να μην είναι πολύ εξελιγμένο το σύστημα, αλλά προσφέρει νομική βεβαιότητα. Επίσης έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει ε, να υπάρχουν κάποια κριτήρια όσον αφορά τους πιστωτές, δηλαδή μπορεί να επιβληθεί ε, και κάποια θυσία σε ε, πιστωτές ασφαλισμένους και μη. Αυτά λειτουργούν πάρα πολύ καλά με μεγάλες εταιρείες. Επίσης έχουμε υιοθετήσει κάποιες δράσεις που αφορούν την αναβολή επιβολής ε, ε, που είναι μόνο για τέσσερις μήνες ε, χωρίς δυνατότητα επέκτωσης. Επίσης είπα, θεωρούμε ότι ήταν καλύτερη μία περίοδος τριών μηνών. Έχουμε και ένα μηχανισμό δεύτερης ευκαιρίας και την προστασία από διαδικασίες αποφυγής, όχι μόνο όταν μιλάμε για νέο χρήμα, αλλά και για οποιαδήποτε αναδιάρθρωση εντός ή εκτός ε, δικαστηρίου. Μια που αναφέρθηκα λοιπόν στο ισπανικό μοντέλο, θα ήθελα να περάσω στο σημερινό μας ε, θέμα. Υποστηρίζουμε πλήρως την προσέγγιση της ε, Κομισιόν και όπως αντιλαμβάνεστε η Ισπανία έχει ευθυγραμμιστεί ήδη πολύ και οπωσδήποτε τα σχετικά μέτρα αυτά θα συνεισφέρουν στο να έχουμε μια ανάκτηση ε, του τραπεζικού χρέους και άρα να μειώσουν το επίπεδο των καθυστερούμενων πληρωμών. Θα ήθελα όμως να σημειώσω κάτι, ότι καμιά φορά θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή έχει εστιάσει υπερβολικά στις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις μικρομεσαίες τουλάχιστον ε, στο μέγεθος που υπάρχει στην Ισπανία. Οι θετικές πτυχές που υπάρχουν και βλέπουμε είναι η εξή. Ε, πρώτα απ' όλα η προστασία του ενδιάμεσου χρήματο κάτι το οποίο θα είναι μια μεγάλη καινοτομία. Αν δεν γνωρίζετε τι είναι αυτό, σημαίνει τα λεφτά τα δίνονται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ενώ τα, το νέο χρήμα είναι το χρήμα το οποίο θα προκύψει από την εκτέλεση της συμφωνίας. Η έννοια λοιπόν αυτή του ενδιάμεσου κεφαλαίου θα είναι μια μεγάλη καινοτομία βεβαίως δεν συμφωνούμε πλήρως με την ανάγκη δικαστικής ε, παρέμβασης. Ε. Πρέπει εδώ πέρα λοιπόν να υπάρχει προστασία ανεξαρτήτως του αν δικασία είναι εντός ή εκτός του δικαστηρίου. Επίσης θεωρούμε ότι η αναβολή εκτέλεσης ε, δηλαδή να δοθεί ένα περιθώριο για να διαπραγματευτεί ο φιλέτης με τους πιστωτές λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Όμως η επέκταση πέρα από τους ε, τέσσερις μήνες θα πρέπει να εξετάζεται μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις και πάντα με βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως παραδείγματο χάρη η στήριξη της πλειοψηφίας των πιστωτών γιατί η τωρινή διατύπωση λέει ότι αν υπάρχει ε, αν υπάρχουν στοιχεία προόδου στι διαπραγματεύσει Είναι πολύ γενικόλογοι. Επίσης, ε, καλοδεχούμενη προσέγγιση των ε, εκτελεστών ε, συμβολέων και συμφωνούμε επίσης στην δυνατότητα να εξαναγκαστούν σε συμβιβασμό οι πιστωτές. Κάτι τέτοιο δεν θα το έλεγα πριν από λίγα χρόνια, αλλά έχοντας την εμπειρία και της σχετικής ε, θυσίας ε, και το όφελος ε, του να μην κλείσουν οριστικά οι εταιρείε πελάτες μας θεωρούμε ότι είναι κάτι το σωστό. Επίσης έχουμε την αρχή ε, ότι δεν θα πρέπει κανένας πιστοτής ε, να ε, βγει σε χειρότερη θέση, δηλαδή να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των πιστωτών, κάτι το οποίο θεωρείται ε, το τεστ για το τι είναι αναλογική θυσία που θα πρέπει να υποστεί ο πιστητής. Τέλος, για τη δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες, το να υπάρχει μια περίοδο απαλλαγής για το χρέος είναι λογικό και για εμάς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γιατί θεωρούμε πως υπάρχει μια κοινωνική ανάγκη, όμως μια ελάχιστη πληρωμή κατά την προηγούμενη περίοδο πρέπει να αξιολογηθεί. Αυτός δεν θα πρέπει να είναι ένας μηχαν... Δεν θα είναι ένας μηχανισμός ε, του να πληρώνει κανείς όποτε μπορεί και βεβαίως υπάρχει και το προαπαιτούμενο της καλής πίστης. Θα μιλάμε για οφειλέτες που λειτουργούν καλή την πίστη και τέλος θα πρέπει να υπάρξει εξαίρεση κάποιων πιστώσεων ε, των δημοσίων παραδείγματο χάρη ε, η οποία όμως περιορίζει τον βασικό στόχο του μηχανισμού δεύτερης ευκαιρίας. Συμπερασματικά Τώρα, όπως σας είπα, εμείς υποστηρίζουμε την πρόταση αυτή. Επίσης θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας ε, που θα τεθούν για να υπάρχουν ε, τα κατάλληλα όρια στους νέους ε, κανόνες. Οπωσδήποτε γνωρίζουμε πως η Κομισιόν αντιμετωπίζει διάφορα μοντέλα εθνικής νομοθεσίας που δύσκολα συμβιβάζονται καθώς βασίζονται σε αντικρουόμενες προσεγγίσεις. Αυτό το οποίο όμως συνέβη τελικά είναι ότι η προτινόμενη οδηγία έχει δανειστεί πολλά χαρακτηριστικά από το κεφάλαιο 11 του αντιστοιχού κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίως ε, διαφέρει πολύ το σύστημά μας από το αμερικανικό. Υπάρχουν λοιπόν δύο βασικά σημεία που θεωρούμε ότι πρέπει να ξαναδούμε στην πρόταση. Το πρώτο είναι ο κανόνας της απολύτου προτεραιότητας ε, όπου δίνεται η δυνατότητα στους ε, πίστοτες ε, να επιβάλλουν σε αυτούς οι οποίοι είναι πιο κάτω στην ιεραρχία να επιβάλλουν την αναδιάρθρωση σε αυτούς οι οποίοι είναι πιο πάνω στην ιεραρχία των πιστωτών. Το πώς θα γίνει αυτό λοιπόν και το πότε βεβαίως δεν είναι σαφές. Θεωρούμε ότι η δυνατότητα αυτή λοιπόν θα πρέπει να απαγορευτεί γιατί θα, έχει την δυνα... θα καταλήξει τελικά στο να μην υπάρχει θέληση να χορηγηθεί η πίστη. Επίσης σχετίζεται με αυτό η διαδικασία ιεραρχίας ε, των πιστωτών. Γιατί εδώ πέρα υπονοείται μια μεγάλη αλλαγή από την νομική βεβαιότητα. Όπως είπα υπάρχουν δύο μόνο κατηγορίες ε, πιστωτών, ασφαλισμένοι και εμεί στην Ισπανία, κάτι το οποίο δημιουργεί νομική βεβαιότητα και έτσι θα πάμε σε ένα σύστημα το οποίο θα εξαρτάται από ιδιωτικές συμβάσεις. Οπότε μπορούμε να αναμένουμε πολύ περισσότερες ε, πρόσφυγες στα δικαστήρια. Και τέλος η δεύτερη καινοτομία αφορά την μεγαλύτερη εμπλοκή των δικαστηρίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κανόνας απόλυτη του προτεραιότητας. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε με την αξιολόγηση ενός ειδικού που θα ορίζει το δικαστήριο ή για την χορήγηση νέας πίστοσης. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, δικαστικός έλεγχος, αλλά πάντα αφού καταλήξουμε σε μια συμφωνία με στόχο να διασφαλίσουμε και τα δικαιώματα του πιστωτή. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελα να σας δώσω σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Ε, αυτά. Ε, thank you very much. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσουμε την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα τον κύριο Λουκ Χέντριξ. UEPMEA, κάπως έτσι. Θα μας πείτε εσείς φαντάζομαι τι είναι ακριβώς το ΕΑΠΜΕ. Α, συγγνώμη, αλλά η κυρία Ρέγνερ έχει μια ερώτηση. Ναι, συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να σας διακόψω. Απλά βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλούς ομιλητές. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και γι' αυτό θέλω να σας παρακαλέσω να πείτε και στους ομιλητές να είναι και αυτοί σύντομοι, να είμαστε και εμείς σύντομοι για να μπορέσουμε να κάνουμε ερωτήσεις, ε, να μην ε, έχουμε μόνο παρουσιάσει. Ναι, πράγματι έχουμε προβλέψει και χρόνο για ερωταπαντήσεις. Ε, ο κύριος Λουκ Χέντριξ λοιπόν τώρα να μας μιλήσει που είναι ο αρμόδιος για την μεταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στις εξωτερικές σχέσεις και τις νομικές υποθέσεις. Δέκα λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Γιούρη που με προσκάλεσε εξ ονόματος της ΟΑΠΜΕ που εκπροσωπεί τους ε, κοινωνικούς εταίρους και τους εργαζομένους. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για τη δουλειά που έχει κάνει. Κύριε Αγκάγιο, αναφέρθηκε και αυτή, ήταν πολύ δύσκολο να συμφιλειωθούν οι διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες ε, με την αυτή πρόταση και ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε τις διαβουλεύσεις με τους εμπλεκομένους φορείς, με την ομάδα τα κτλ. πραγματικά ήταν πάρα πολύ θετική. Και λοιπόν η πρόταση γίνει ισορροπημένη. Με αυτή την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια νέα προσέγγιση για τα θέματα της αφαιρεγκαιότητας επί οδηγία solvency ε, πιο ε, εκτεταμένη από την αρχική πρόταση του 2014 που δεν έχει εγκριθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η πρόταση δεν έχει στόχο να εναρμονίσει κάποιες βασικές πτυχές της αφαιρεγγιότητας, όπως είναι οι όρκοι προϋποθέσεις για την κίνηση διαδικασίων αφαιρεγγιότητας, κοινορισμό ή κατάταξη των απαιτήσεων και δράσης αποφυγής κτλ. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι θα ήταν κάτι τέτοιο πάρα πολύ δύσκολο, και αδύνατο για την εναρμόνιση δηλαδή κατηγοριών πιστωτών. Βέβαια, πρέπει να πω ότι επειδή οι πιστωτές ε, είναι εκτεθειμένοι σε διάφορους κινδύνους ε, και αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση ε, και να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφορες διεκδικήσεις. Θα κάνω κάποιες γενικές παρατήσεις και μετά κάποιες πιο εξειδικευμένες παρατήσεις. Στόχος της Κομισιόν είναι ε, η πρόορη αναδιάρθρωση του χρέου για προστασία των θέσεων εργασία και πρόθεση τη ανάπτυξη. Και αυτό μπορούμε νομίζω να το υποστηρίξουμε γιατί πάρα πολλέ επιχειρήσει πτωχεύουν ετησίω. Ένα από του σημαντικότερου στόχου αυτή τη πρόταση είναι να υπάρχει αυτή η νοοτροπία ε, για διάσωση, για επιβίωση της επιχείρησης. Και αν αυτό δεν είναι δυνατό να υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία καθάρισης. Στο πλαίσιο της πρότασης ε, έχει να κάνει ακριβώ και με τα ποσοστά ανάκτησης ε, των δανείων των πιστωτών. Επίσης, δεύτερη ευκαιρία που δίνεται στους έντιμους ε, επιχειρηματίες. Εάν δηλαδή αποτύχει μια επιχείρηση, ο επιχειρηματίας μπορεί να αποσβέσει το χρέος του σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και να έχει τη δυνατότητα επίσης να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, να ξεκινήσει μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα παρά την αποτυχία την πρώτη. Αφαιρεγγιότητα δηλαδή δεν θα πρέπει να οδηγεί σε κοινωνική ή και οικονομική στιγμα... σε κοινωνικό στιγματισμό ή οικονομικό στιγματισμό ε, και θα πρέπει να προωθείται η οικονομική βιωσιμότητα και ανάκτηση των κονδυλίων των ψητών. Θα πρέπει λοιπόν να τις προσεγγίσει να στηρίζεται η ανάπτυξη, η επιχειρηματικότητα και η απασχόληση. Δεν θα πρέπει να χαθούν θέσει εργασία ή επιχειρήσει λόγω των πτωχεύσεων. Αν όμω ο επιχειρηματία αποτυγχάνει από οικονομική και κοινωνική πλευρά, είναι σωστό και δίκαιο το άτομο αυτό να μπορεί να κάνει μια καινούργια αρχή το στομότερο δυνατό. Για να πετύχουμε λοιπόν ένα κατάλληλο πλαίσιο αφαιρεγγιότητα, εμεί θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα, να βρεθούν τι βιώσιμε επιχειρήσει να μπουν στην ε, διαδικασία αναδιάρθρωση. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρωταρχικό μέλημα στι δικασίε αφαιρεγκαιότητα. Είναι και σημαντικότερε. Με την προπόθεση ότι η επιχείρηση είναι βιώσιμη. Οπότε τότε μια επιχείρηση που αντιμετωπίζει δυσκολίε θα πρέπει να μπορεί να εντοπιστεί εγκαίρω και να τη προσφερθούν οι, ε, η απαιτούμενη βοήθεια και υπό τη μορφή της αναδιάρθρωσης. Όμως ο στόχος του προληπτικού μέτρου είναι να εστιάζει σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσκολία. Και μπορούν όμως να βοηθηθούν χωρίς να χρειάζονται μέτρα αναδιάρθρωσης που είναι και μακροχρόνια και δαπανηρά. Αν λοιπόν δεν χρειάζεται η αναδιάρθρωση, μειώνεται ο αντίκτυπος στους πιστωτές και στους εργαζόμενους. Αν χρειαστεί αναδιάρθρωση θα πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της επιβίωσης της επιχείρησης αφενός και των δικαιωμάτων των πιστωτών αφετέρου. Θεωρούμε λοιπόν εν γέννη την πρόταση ως θετική, περιλαμβάνει κατά την άποψή μας μια καλή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των πιστωτών και των σφαιρόντων των ε, δανειζομένων. Βέβαια υπάρχουν κάποια θέματα όπως ε, η προληπτική αναδιάρθρωση. Όταν μιλάμε για προληπτική αναδιάρθρωση, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να φροντίζουν τα δικαιώματα των πιστωτών να προστατεύονται επαρκώς, ιδίως αν χρειαστεί να υπάρξουν μεμονωμένες διαταγές ε, εκτελέσεις και οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν τους πιστωτές οπότε ο κατάλογος των πιστωτών τα μέτρα που θέλει να πάρει ο, φιλο, ο φιλέτης όλα αυτά θα πρέπει να δίνονται ε, σε δικαστή ε, για να έχει ενημέρωση εκ των προτέρων και θέλουμε αυτό να αναφέρεται στην πρόταση. Και θα κάνουμε και μια συγκεκριμένη τροπολογία. Σε ό,τι αφορά αυτό το τίτλο για να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες, ε, τους έντιμους επιχειρηματίες. Πράγματι, η, δεύτερη ευκαιρία είναι το θέμα. Εταιρείε, ενώσεις. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα απαλλαγής. Μέσα σε τρία χρόνια την έναρξη της διαδικασίας αφαιρεγγιώτες. Είναι μεν αυτή η πρόταση και αυτό το σχέδιο αναδιάρθρωσης μια καλή ε, αρχή, αλλά πρέπει να είναι οριστικές προθεσμίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί μπορεί να μην επιτευχθεί με βάση εθνικές προθεσμίες μια συμφωνία. Άρα η δεύτερη ευκαιρία θα είναι υποκειμενική και όχι αντικειμενική. Θεωρούμε ότι είναι θεμητό να υπάρξει μια, μια δεσμευτική προθεσμία όταν έχουμε να κάνουμε έναν έντιμο επιχειρηματία. Όμω λέει το άρθρο 20, θα πρέπει να δοθεί απαλλαγή μέσα σε τρία χρόνια. Για τι περισσότερε ε, περιπτώσει τα μέλη μα θεωρούν ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί αν ο φιλέτη είναι μη συνήθω οι διαδικασίε είναι απλέ. Άρα η αρχή είναι ότι όταν μιλάμε για έναν έντιμο επιχειρηματία, θα πρέπει η απαλλαγή να γίνεται μέσα σε ένα έτό από την έναρξη τη διαδικασία περιγκαιότητα. Εκτό αν είναι πιο πολύπλοκη υπόθεση με βάση το δικαστήριο οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί δεν συμφωνούν με το ένα έτος, πρέπει να σας πω, ούτε και με τα τρία χρόνια. Και απλά και θα πρέπει να γίνεται μόνο μετά από πρόχευση και αν έχουμε διαδικασία αναδιάρθρωσης η απαλλαγή θα πρέπει να δίνεται μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Έπειτα έχουμε μια συγκεκριμένη τροπολογία ότι η απαλλαγή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για έντιμους επιχειρηματίες και νομίζω το πήκε η κυρία Γκάιο. Άρθρο 20. Θα πρέπει λοιπόν να, τροπολογήσουμε τροποποιηθεί αυτό το άρθρο προ αυτή την κατεύθυνση. Θα επιμείνουμε όμω και ακόμα πιο, πιο μακριά σε ό,τι αφορά το τεκμήριο τη εντυμότητα του επιχειρηματία. Σε ό,τι αφορά δηλαδή, την αντιστροφή του βάρου απόδειξη. Στο τίτλο 4 για τα μέτρα βελτίωση αποτελεσματικότητα αναδιάρθρωση. Εδώ η πρόταση έχει ω ως στόχο για αναδιάρθρωση και η περιγκαιότητα ω διαδικασίε να είναι πιο αποτελεσματικέ πιο ταχείες και πιο απλές. Πιο σύντομες με λιγότερο κόστος, γιατί αυτό είναι προς το οικονομικό όφελος και των φιλετών και των πιστωτών. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Καλώς ορίζουμε την πρόταση αυτή για την υποχρέωση που έχουν τα κράτη-μέλη από αυτού. Σε ό,τι αφορά τα διάφορα μεγέθη επιχειρήσεων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες τους ε, αναλόγως. Η αναδιάρθρωση πρέπει να είναι δυνατή για όλες τις επιχειρήσεις, σε οδήποτε μεγέθους. Αλλά για κάποιες επιχειρήσεις είναι και ε, δύσκολο και πολύ δαπανηρό. Πάνω για μια μικρή κλίμακα επιχείρηση. Η διάρκεια μπορεί να είναι επίση μεγάλη, μπορεί να χρειαστεί ένα χρόνο από την αίτηση μέχρι την επιβεβαίωση, την έγκριση του σχεδίου. Και επειδή έχουν δημιουργηθεί νέε θέσει εργασία τα πρόσφατα χρόνια, ιδίω από ΜΜΕ, η αναδιάρθρωση, ξέρουμε ότι θα πρέπει να είναι μια βιώσιμη επιλογή και για αυτέ τι επιχειρήσει και η αρχή του first ε, come, first serve πρέπει να λέμε την υπόψη. Τέλος. Θέλω να σας θυμίσω τις προτάσεις που έχουν ήδη γίνει και συμφωνηθεί στο Small Business Act. Και έχει εγκριθεί από τα κράτη-μέλη αυτή η νομική πράξη και από την Κομισιόν ήδη από το 2008. Εκεί λοιπόν 2008 δηλαδή λεγόταν ότι θα πρέπει τα κρατημένα να φροντίσουν οι έντιμοι επιχειρηματίε που αντιμετωπίζουν το φάσμα τη πτώχευση να μπορούν να έχουν γρήγορα μια δεύτερη ευκαιρία και ότι τα κράτη-μέλη επίση καλούνται να προωθήσουν μια θετική στάση στην κοινωνία για να μπορεί να δοθεί μια νέα αρχή σε αυτού του επιχειρηματίε, ό,τι αφορά πριν χάρη δημόσιε ενημέρωση. Και επίση ότι όλε οι νομικέ διαδικασίε για την καθάριση αν δεν υπάρχει δόλια, τα όχι πρέπει να ολοκληρώνονται μέσα σε ένα χρόνο και η επανεξα... επανέναξη θα πρέπει να υποστηρίζεται. Αυτά τα συμφώνησαν τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν το 2008. Νομίζουμε ότι αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν και σε αυτήν την οδηγία. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι έμεινα και στο δεκάλεπτο που μου είχατε δώσει. Ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστούμε. Τώρα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και την οπτική τους γωνία ο κ. Πέτερ Σέρερ, αναπληρωτής γενικός γραμματής της ETUC, γνωστής και ως ΕΤΟΚ. Έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα κάνω την παρουσίασή μου ε, στην ε, λογική γενικών παρατηρήσεων και κάποιων συγκεκριμένων συστάσεων. Η αναθεώρηση του νόμου περί είναι πολύ σημαντική για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ιδίως σε καιρούς κρίσης, όπου οι εργαζόμενοι έχουν ε, την αίσθηση ότι κανόνες περί τους ε, πλήττουν άμεσα με απολύσεις χωρίς πρώτερη προειδοποίηση, με μη πληρωμή μισθών και αμοιβών ή άλλων δικαιωμάτων που τους αναλογούν. Η επικέντρωση τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να είναι οι τράπεζε και η υποτεμισιακή του μεταχείριση, αλλά η προστασία των εργαζομένων στην αναδιόρθρωση και τι περιπτώσει αφαιρεγγιότητα. Η πρόταση πρέπει να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη χρήση των τακτικών αφαιρεγγιότητα, που όλο ένα και χρησιμοποιούνται περισσότερο, για να διαφεύγει κανεί των ευθυνών του από όσα προκύπτουν από το, εργατικό δίκαιο και το αστικό δίκαιο και γι' αυτό βλέπουμε και σκάνδαλα να έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια ε, προκαλώντα προβλήματα σε χιλιάδες εργαζομένους και με μεγάλο κόστος για τεχνικά συστήματα κοινωνική ασφάλεια, όπως η Αλιτάλια, η έστρο στι ε, κάτω χώρε, που ε, άφησε άνεργου χιλιάδες εργαζομένους και για του εναπομείνοντε εργαζομένου προέβλεψε κάκιστες συνθήκες εργασίας. Το ίδιο και όλε οι, ε, οι εξετασμένε ήδη αξιώσει. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν ε, του μισθού και τι αμοιβέ του ε, άμεσα και χωρί καθυστέρηση. Θα πρέπει επίση να έχουν το καθεστώ του προτιμησιακού δανειζόμενου, όσο και αν το ασφαλιστικό σύστημα αυτή τη στιγμή πλήττεται από τις προτάσεις περί οι εργαζόμενοι είναι μια ξεχωριστή κατηγορία από μόνοι του. Οι νόμοι σκοπεύουν να σώσουν τι επιχειρήσει και τι θέσει εργασία, αλλά θα πρέπει να υπάρχει πλήρη ενημέρωση, διαβούλευση και συμφωνία με του εργαζομένου και του εκπροσώπου του. Η στήριξη για κάθε νέο ε, κανονισμό σε επίπεδο οργανισμού είναι σημαντική. Ε, η αναδιάρθρωση του χρέους όπως ο ονομαστή διασταυρούμενης τάξης και κατηγορίας έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους εργαζομένους και πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς ε, εγγύησεις. Θα πρέπει να υπάρξει βιωσιμότερη και υπευθυνότερη επιχειρησιακή συμπεριφορά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε οι εταιρείε να σέβονται τα συμβασιακά τους καθήκοντα λαμβάνοντας υπόψη τις πρακτικές και τους νόμους που ισχύουν και για τους ίδιους και για τους εργαζομένους ε, αλλά το ίδιο και οι νομικοί εμπειρογνώμονε για να προστατευόμαστε από τι παραβιάσει. Ε, ο στόχο τη προστασία των θέσεων εργασία είναι το πλέον σημαντικό για μα. Ε, ενώ τα σχέδια αναδιάρθρωση έχουν σοβαρέ επιπτώσει στον χώρο εργασία στι συμβάσει πρόσληψη και στι συλλογικέ διαπραγματεύσει, η προτινόμενη οδηγία θα πρέπει να διασφαλίσει ρητό τα δικαιώματα των εργαζομένων στην ενημέρωση, διαβούλευση και συμφωνία σε όλε τι φάσει τη διαδικασία δεν αρκεί απλώς να δηλώνεται ότι η οδηγία επιφυλάσσεται των συμπεφωνημένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, διαθετήσεων για την ενημέρωση και τη διαβούλευση. Πρέπει ο Ευρωπαϊκός Νομοθέτης να βεβαιωθεί ότι υπάρχει ε, βιώσιμη και για όλους διαδικασία, μεταξύ των οποίων ε, θα πρέπει να περιλαμβάνει την υποχρέωση αυτό που διοργανώνει την ε, αναδιάρθρωση να ενημερώνει όλους όσοι θα επηρεαστούν ε, στην θέση απασχόλησής τους, στη δουλειά τους και θα επηρεαστούν και τα δικαιώματά τους, ότι η εταιρεία πρόκειται να πτωχεύσει. Η ιδέα αυτή θα πρέπει να προσθεθεί στα άρθρα 8 και 9. Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που θα πλήξει το μισθολόγιο και τις εργασιακές συνθήκες δεν μπορεί να γίνει νομικός δεσμευτικό απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης και συμφωνίας με τους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με τους εκπροσώπους τους θα πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν εναλλακτικά σχέδια αναδιαρθρωσής για να προστατεύσουν θέσεις εργασίας βάσει ε, εξωτερικής εμπορογνωμοσύνης ε, για αντιπροτάσει. Αυτό θα πρέπει να προσταθεί στο άρθρο 9. Η οδηγία πρέπει να βεβαιωθεί ότι τα εργαλεία έγκαιρη προειδοποίηση που διατίθενται στι επιχειρήσει είναι γνωστά και στου εκπροσώπου των εργαζομένων. Γι' αυτό ζητούμε μια προσθήκη για το θέμα αυτό στο άρθρο 3. Η οδηγία πρέπει να προσφέρει βεβαιότητα ως προς την ανάγκη να γίνονται οι σεβαστά τα συστήματα κανονικών ή μηχανικών επιχειρησιακών σχέσεων. Αυτό μπορεί να γίνει στο άρθρο 31. Η οδηγία πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων να προστατεύουν τα δικά του συμφέροντα μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών δράσεων, μεταξύ των οποίων η απεργία βάσει και του άρθρου 27 και 28 της Χάρτας των Θεμελιδών Δικαιωμάτων αυτό θα πρέπει να αναφέρονται στα άρθρα 9, 11 και 31 της προτινόμενης οδηγίας. Η οδηγία πρέπει να βεβαιώνεται ότι τα συνταξιδοτικά ταμεία δεν πλήττονται και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στο άρθρο 9 θα πρέπει να υπάρχει πλήρη δέσμευση για την προστασία των συνθηκών εργασία των εργαζομένων πριν τη διαδικασία αναδιάρθρωση. Η ΕΤΟΚ προτείνει ένα νέο άρθρο 12B, 12α, το οποίο μπορεί να προσθεθεί στο σχέδιο του κειμένου ε, για να συμπληρώσει τα σημεία που λείπουν. Τα κράτη-μέλη τα κράτη θα πρέπει να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία τη αναδιάρθρωση, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα των εργαζομένων στι συλλογικέ διαπραγματεύσει, τη συλλογική δράση ε, και το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη διαβούλευση ενημέρωση για κάθε στοιχείο που μπορεί να προκύψει και να πλήξει την απασχόληση και την απασχολησιμότητα των εργαζομένων ε, ή τουλάχιστον να πάρουν τους μισθούς που τους αναλογούν. Ε, ορκωτό με λογιστικό έλεγχο ε, πρώτης διαδικασίας αναδιάρθρωσης και προτιμησιακή μεταχείριση των εργαζομένων ως δανειζομένων. Θα πρέπει τα κατημελή να βεβαιωθούν ότι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ξεχωριστή κατηγορία από μόνοι του και οι μισθοί αλλά και οι θέσει απασχόλησή του λαμβάνονται υπόψη και σε περιπτώσει αναδιάρθρωση και πτώχευση. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να διασφαλιστούν οι αξιώσει των εργαζομένων, η κατηγοριοποίησή του ω ασφαλών και προτιμησιακών δανειζομένων, κάτι που δεν μπορεί να ε, αμφισβητείται, και να ε, υποβιβαστεί από οποιονδήποτε άλλο δανειστή. Είναι ξεχωριστή κατηγορία, αυτό θα πρέπει υποχρεωτικώ να αναγνωρίζεται και να αναφέρεται στο άρθρο 12α. Εάν δεν ισχύσουν όλα αυτά, θα πρέπει μια εταιρεία να αναστέλει τη δράση της. Δεν μπορεί οι εργαζόμενοι να χάνουν μισθούς, να μην έχουν γνώση ή να χάνουν τα δικαιώματά τους, τις διακοπές τους, τις συντάξεις τους, τα μπόνους τους. Ό,τι του αναλογεί ανάλογα με την εργασιακή σχέση που είχε διαμορφωθεί με την εταιρεία. Προτείνουμε λοιπόν αλλαγέ στο άρθρο 6 που να βεβαιώνουν ότι οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν όλα τα δικαιώματα πλήρω και χωρίς καθυστερήσεις περιορίζοντας την προθεσμία των 70, στις 70 ημέρες μαζί με τις παρατάσεις και τις ε, ανανεώσεις. Όλα αυτά θα πρέπει να ξεπερνούν τις 100 μέρες στη χειρότερη περίπτωση και θα πρέπει να διασφαλιστούν και σαν προβλέπει η Οδηγία 9859 ΕΚ ε για τις συλλογικέ απολύσεις και η Οδηγία 2001-23 που ε, προβλέπει τους όρους για την πρόσληψη σε περίπτωση μεταφοράς εταιρεία κατά τη διάρκεια διαδικασίας πτώχευσης. Εκεί χρειάζεται αλλαγή στο άρθρο 1. Το να έχουμε πιο βιώσιμη εταιρική συμπεριφορά, ε, κατά την άποψη της ΕΤΟΚ, έχει να κάνει με τους κανόνες που θα προσφερθούν για να υπάρχει μια δεύτερη ευκαιρία. Όμως δεν είναι βέβαιο ότι οι ελεγκτές μια εταιρεία και οι λογιστές της ε, όταν κοιτάζουν την αφαιρεγιότητά της λόγω δική τη ε, κακοδιαχείρισης ειδικών τη ευθυνών, θα πρέπει να τους συγχωρεί από κάθε χρέος και δανειοδότηση. Θα πρέπει να μην τους δίνεται το προνόμιο της περιορισμένης ευθύνης. Οι εταιρείε αυτές δεν θα πρέπει να μπορούν να παρακάμπτουν το εργασιακό δίκαιο, να περνάνε σε αθέμητο ανταγωνισμό και να συμπεριφέρονται κοινωνικά ανεύθυνα. Αυτά πρέπει να αναφέρονται στα άρθρα 19 και 22 οι διευθυντέ, οι επιχειρηματίε και όσοι είναι υπεύθυνοι για τι διαδικασίε πτώχευση πρέπει να λογοδοτούν και να υπάρξει αποτρεπτική ε, πρόβλεψη στον νόμο για να είμαστε σίγουροι ότι προστατεύονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η ΕΤΟΚ πιστεύει ότι υπάρχει περιθώριο ελπίδα στα άρθρα 19, 21, 22, 23 και 25. Και ναι, το συμπέρασμά μου συνολικά είναι, όπως είπα ευθύς εξ αρχής, ότι την πρόταση αυτή την κοιτάμε από την προοπτική των εργαζομένων και όχι μόνο των τραπεζών και των κεφαλαιοκρατών. Θέλουμε να προστατεύσουμε του μισθού και τα δικαιώματα των εργαζομένων, τα δικαιώματα στην ενημέρωση και τη διαβούλευση και το δικαίωμα στι συλλογικέ διαπραγματεύσει και τη συλλογική δράση. Αυτά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραβιάζονται. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσουμε την άποψη των ατόμων που δραστηριοποιούνται επί τόπου στο θέμα. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Άξελ Μπίρμπαχ από την Γερμανία για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Νίμπλερ, κυρίες και κύριοι, ασχολούμαστε εδώ και 20 χρόνια με επιχειρήσεις κρίση στην ε, Ένωση ΦΕΟ ή ΔΕ την Ένωση διαδικασιών αφαιρεγγιότητας. Έχουμε 470 μέλη που είμαστε όλοι επαγγελματίες διαχειριστές και υποστηρίζουμε την πρόταση αυτή οδηγίας και τον στόχο της για να διευκολύνει την αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων. Αλλά η εμπειρία μας με την συμπεριφορά επιχειρήσεων στην κρίση και των πιστωτών σε καταστάσεις κρίσης μας αρέσει να βλέπουμε πάρα πολύ ε, επικριτικά κάποιες προτάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ και σε κάποιους ε, κινδύνους που αφορούν τη γενικότερη οικονομία, την μακροοικονομία. Η Ένωσή μας ε, θεωρεί πως ε, υπάρχουν πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Οι σημαντικότερες λοιπόν από αυτές είναι αυτές που αναφέρω τώρα. Πρώτα απ' όλα περιοριζόμαστε στους ε, πιστωτές που είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι δύο στόχοι δηλαδή που είναι αφενός ε, να ελαφρύνουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υψηλό χρέος αλλά είναι βιώσιμες και από την άλλη να αναδιαρθρωθούν τα μη ε, εξυπηρετούμενα δάνεια μπορούν να εξυπηρετηθούν με απλούστερους ε, τρόπους. Η δημιουργία ε, ενός περιορισμένου μη γραφειοκρατικού και αποτελεσματικού συστήματος νομίζω πως επαρκεί για να αποφύγουμε επίσης κινδύνους στην μακροοικονομία, στη γενικότερη οικονομία θα μπορούσαμε να δούμε πόσο θα αποφύγουν τον κίνδυνο οι προμηθευτές και οι λυπήπιστετές. Επίσης η πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη που θα σημάνει αυτό σε αλλαγή του εργατικού δικαίου, του εταιρικού δικαίου και του φορολογικού δικαίου μπορεί να αποφευχθεί. Δεύτερον, θα οδηγηθούμε σε πιο ακριβή πίστοση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η οδηγία αυτή αντιτίθεται στο άρθρο 178 της Οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων. Γιατί αναγνωρίζετε πως ε, υπάρχει η δυνατότητα εξασφάλισης ε, μετά από 90 μέρες όταν πλέον δεν έχει το δικαίωμα ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να εκποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Ε, θα μπορούσε λοιπόν πάρα πολύ σύντομα μετά το μοτατόριο σύμφωνα με το άρθρο 6 και 7 να οδηγηθούμε σε ένα α, στον χαρακτηρισμό ενός δανείου μη εξυπηρετούμενο σύμφωνα με την οδηγία CRR. Θεωρούμε λοιπόν πως ε, το μορατόριο 4 μηνών είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον αυξάνει την πίεση στο ίδιο κεφάλαιο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ε, χορήγηση δανείων, κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κόστος του χρήματος. Επίσης, ανισχυτικό είναι το ότι η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων θα μπορούσε τελικά να μεταφερθεί σε μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα μικρότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εάν δεν έχουν, ε, αν δεν οδηγηθούν σε μια αύξηση του κόστους ε, του χρήματος, ε, θα αναγκαστούν να χωριστούν από πάρα πολύ πάρα πελάτες τους, οι οποίοι κατά κύριο λόγο βέβαια βρίσκονται στην ε, περιφέρεια. Τρίτον, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος ε, επακόλουθων χρεοκοπιών. Η πιθανή συμπερίληψη όλων των πιστωτών στο ε, προγραμματισμένο αυτό μορατόριουμ αποτελεί κίνδυνο για τους προμηθευτές των επιχειρήσεων συχνά μιλάμε για περιθώρια πληρωμών 60, 90 ή και 180 ημερών, κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι προμηθευτές με θα κινδυνεύουν με χρεοκοπία οι ίδιοι. Μία αναβολή λοιπόν των μέτρων εκτέλεσης, στο μορατόριουμ το οποίο προτείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 και 7 της ε, οδηγίας ε, σημαίνει ότι θα υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες παρατάσεις ε, των προθεσμιών πληρωμός και άρα έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος μη πληρωμής, κάτι το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο για τους προμηθευτές. Και δεν πρέπει εδώ πέρα να παραβλέπουμε ότι συχνά και οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να αγοράσουν μεγάλα και ακριβά τμήματα του ίδιου του προϊόντος. Οπότε οι απαιτήσει αυτές σημαίνει ότι τελικά θα οδηγηθούμε στο ότι δεν θα δέχονται τις εγγυήσεις αυτών των επιχειρήσεων των προμηθευτών ή τράπεζες και εταιρείε factoring. Τέλος, δεν υπάρχουν, ε, άρα δεν υπάρχει αρκετό ρευστό σε κλάδους όπως παραδείγματο χάρη οι προμηθευτές των αυτοκινητοβιομηχανιών ή ο κλάδος των ε, τροφίμων. Οι προτάσεις αυτές λοιπόν θα λειτουργήσουν ε, μόνο εις, βάρος των χρε... εις ε, όφελος των χρεωμένων επιχειρήσεων ε, και όχι υπέρ των πιστωτών, κάτι το οποίο δεν είναι αναλογικό. Επιπλέον φοβούμαστε ότι οι πιο ενημερωμένοι εκ των ε, πιστωτών που διαπραγματεύονται με τις επιχειρήσεις θα μπορέσουν να οβεληθούν εις βάρος αυτών οι οποίοι δεν έχουν αυτήν την ενημέρωση. Στην περίπτωση λοιπόν της πτώχευσης μιας ε, επιχείρησης υπάρχει ο κίνδυνος ο οποίος αυξάνεται περισσότερο για αυτούς οι οποίοι θα έχουν υποστεί το μορατόριο. Μπορεί λοιπόν να περιοριστεί αυτός ο κίνδυνος μέσω μιας ε, ανεξάρτητης, ενός ανεξάρτητου τρίτου διαχειριστή. Ήδη σήμερα βλέπουμε πως ε, η εμπιστοσύνη συχνά ε, υπάρχει μόνο σε ε, διαχειριστές οι οποίοι έχουν οριστεί από το δικαστήριο. Επίσης υπάρχει, θα δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα φέρει σε πολύ μειονεκτική θέση τους πιστωτές σε σχέση με τους εργαζόμενους, τους μετόχους ε, της επιχείρησης ε, και τους προμηθευτές τους. Και οι κίνδυνοι βεβαίως θα πρέπει να μπορούν να μοιραστούν ε, ισορροπημένα στην αγορά. Χωρίς έναν ουσιαστικό κίνδυνο χρεοκοπίας υπάρχει ηθικός κίνδυνος. Θα πρέπει να έχουν και έχουν βεβαίως υψηλότερο κίνδυνο οι επιχειρηματίες. Το να μην υπάρχουν λοιπόν οι υποχρεώσεις ε, αυτές ε, της χρεοκοπίας σημαίνει ότι θα έχουμε μια κατάχρηση του συστήματος. Η οδηγία αυτή θα πρέπει να σκοπεύει αποκλειστικά στην προστασία, φαίνεται ότι σκοπεύει αποκλειστικά στην προστασία των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, έτσι όμως κινδυνεύουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντος. Δεν υπάρχουν επίσης ξεκάθαρες προϋποθέσεις ε, πρόσβασης μέχρι σε ποιο στάδιο μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την πρόταση η επιχείρηση. Υπάρχει έλλειψη ενός διαχωρισμού από την ουσιαστική χρεοκοπία. Και έτσι κινδυνεύουν οι πιστωτές, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές μιας επιχείρησης, αλλά και οι αγορές συνολικά θα πρέπει να προστατευτούν από μια επιχείρηση η οποία θεωρητικά έχει περάσει μια φάση αναδιάρθρωσης αλλά στην πράξη ουσιαστικά έχει χρεοκοπήσει. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη τρίτη εξέταση της ε, κάθε περίπτωσης ε. κατά τη διάρκεια αυτής ε, της διαδικασίας δεν εξετάζεται καμία απέτηση. Και βεβαίως πιθανές ε, χειραγωγήσεις ε, εδώ πέρα ευνοούνται από αυτό το σύστημα για γνωστούς ε, και φίλους του επιχειρηματία οι οποίοι μπορεί να εκμεταλλευτούν την κατάσταση την στάση δηλαδή πληρωμών έναντι των πιστωτών. Ειδικά οι μικροί πιστωτές δεν μπορούν να προστατευτούν από μια τέτοια χειραγώγηση. Γάμα. Η πρόταση αφήνει ανοιχτό περιθώριο στα κράτη-μέλη το ε, να κρίνουν εάν θα πρέπει να υποβάλει η επιχείρηση μία αίτηση χρεοκοπίας. Οι πιστωτές όμως δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2. Οι πιστωτές δεν μπορούν να εμποδίσουν την διαδικασία αναδιάρθρωσης μέσω κάποιας δικής τους αίτησης ανακοπής. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια εποπτεία του ε, οφειλέτη θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια διαδικασία εκπροσώπησης ε, των συμφερόντων των πιστωτών. 4. Η πλειοψηφία για την ε, ψηφοφορία για την έγκριση ενός τέτοιου σχεδίου αναδιάρθρωσης είναι σύμφωνα με την πρόταση οδηγίας 75% ανά ομάδα πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 9 παραγραφός 4. Ε, Αυτό οδηγεί στον κίνδυνο να επικρατήσουν τέτοιες ε, διαδικασίες φοφορίας επενδυτών που δεν έχουν στρατηγικό συμφέρον. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα χειραγώγησης κάποιων απαιτήσεων. Ε, η πρόταση οδηγία προβλέπει στο άρθρο 17 κατά τη διάρκεια του μορατόριου αυτού να ληφθούν μέτρα προστασίας. Όλες οι συνήθεις ε, πληρωμές ε, της ε, επιχείρησης η οποία είναι οφειλέτης αλλά και μεταβολές κεφαλαίου όλα αυτά σταματούν. Αυτό ουσιαστικά είναι πρόσκληση για κατάχρηση συστήματος. Θα πρέπει η διαδικασία αυτή να μην μπορεί να δίνει την ευκαιρία στο να φύγουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία από την επιχείρηση. Τελευταίο σημείο, βλέπουμε πως ε, παρόλες τις ε, ζημίες δεν αναγκάζεται μια εταιρεία να χρεοκοπήσει και να βγει από την αγορά. Τι σημαίνει αυτό ότι οι επιτυχείς εταιρείε είναι αναγκασμένες να μπορέσουν να, χρηματοδοτούν τις ε, εταιρείε οι οποίες δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν το χρέος τους. Ε, οι προμηθευτές και οι πελάτες, αλλά και οι εργαζόμενοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην επιχείρηση αυτή και στην χρεοκοπία η οποία θα ακολουθήσει τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Uh, ευχαριστώ πολύ και τώρα η δεύτερη προοπτική από έναν επαγγελματία η κυρία Βαλερή Λελούπ από τη Γαλλία έχει το λόγο για δύο, δέκα λεπτά. Merci, Monsieur le Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί έχετε καλέσει και τους επαγγελματίες, ε, τους Γάλλους, ε, επαγγελματίες που έρχονται στον κλάδο των αναδιορθώσεων. Πρέπει να σας πω ότι μας ε, ενθουσίασε η πρόταση της οδηγίας ε, είναι η γαλλική μας πλευρά αυτή. Βέβαια, έχουμε και κάποιες κριτικές να εκφράσουμε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας επενθυμίσω ότι στη Γαλλία επαγγελματίε της αφαιρεγγιότητας χωρίζονται σε δύο ε, επαγγέλματα. Έχουμε τους κατεπάγγελμα συνδίκους και τους διαχειριστές. Οι σύνδικοι παρουσιάζουν το σχέδιο και οι διαχειριστές βλέπουν και, το τη συλλογική διαπραγμάτευση και προσπαθούν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση για την εκαθάριση του παθητικού και για να συνεχίσει η εταιρεία τη δραστηριότητα. Έχουμε έναν ε, σύνδικο μαζί μας, ε, η κυρία εδώ, και αν θέλει απαντήσει, ε, αν θέλετε μπορείτε να απαντήσει. Η τελευταία μεταρρύθμιση με τον νόμο Μακρόν προβλέπει ότι πέραν των επαγγελματιών, αυτών δηλαδή που είναι γραμμένοι στους εθνικούς καταλόγους, έχουμε και τους επιμελητές και τους δημοπράτες που μπορούν να αναλάβουν τις συλλογέ διαδικασίες στη Γαλλία σε ό,τι αφορά μικρές δικαστικές εκαθαρίσεις. Μικρές, δεν είναι καθόλου μειωτικό. Απλά μιλώ για διαδικασίες που γίνονται πολύ γρήγορα γιατί έχει μικρό ε, ενεργητικό και δεν έχει παραλίγους μισθωτούς επιχείρηση. Το ε, δικαστήριο τώρα θα ορίσει ή και σύνδικο και ε, διαχειριστή για όλα αυτά τα θέματα. Εμάς, το επάγγελμά μας είναι νομικός κατοχυρωμένο. Έχουμε 430 επιτελματές, 126 είναι οι σύνδικοι και 304 είναι οι διαχειριστές. Ε, και υπάρχει μεγάλος ε, έλεγχος όσον αφορά το, την πρόσβαση. Υπάρχουν δύο εξετάσεις ε, πάρα πολύ πολύπλοκες που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει κανείς. Θέλει να έχει πραγματικά πολύ μεγάλες δεξιότητες και πολλά προσόντα, χωρίς να θέλω να περιευτολογήσω. Η προσέγγιση τώρα, θέλω να σας δείξω από τη γαλλική σκοπιά πώς βλέπουμε τα πράγματα. Θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις που μπορούν πολύ εύκολα να μεταφερθούν στο εσωτερικό δίκαιο, ενώ άλλες όχι τόσο και θα, για αυτές θα χρειαστούν κάποιες προσαρμογές. Δεν ξέρω μάλιστα μήπως κάποιες φορές υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Σε ό,τι αφορά τα θετικά στο γαλλικό δίκαιο ήδη υπάρχουν πολύ σημαντικά εργαλεία τα οποία συνάδουν με ορισμένες από τις ε, απαιτήσει που θέτει η πρόταση οδηγία ε, δεν θα είμαι διεξοδική γιατί μας μετράτε εδώ πέρα και τα λεπτά, αλλά να σας πω ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τον πρώτο άξονα της πρότασης, μπορούμε να πούμε ότι η χρήση των προληπτικών διαδικασιών είναι κάτι ήδη γνωστό στη Γαλλία, επειδή έχουμε ήδη τη διαδικασία της προειδοποίησης, του εγκαίρου συναγερμού, πρέπει να σας πω ότι οι ελεγκτές έχουν, αυτό το, έχουν αυτή τη δυνατότητα ε, να κρούν τον κόδωνα του συναγερμού και υπάρχει ε, και από το εμποροδικείο μια σχετική διάταξη που προβλέπει ότι αν ε, υπάρχουν προνομιακές εγγραφές σε μια επιχείρηση ε, ο δικαστής, ο αρμόδιος, ε, επιλαμβάνεται για να δει κατά πόσον πρέπει να ξεκινήσει μια συλλογική διαδικασία ή μια προληπτική διαδικασία και κατά πόσον υπάρχουν κάποιοι προνομιακοί πιστωτές. Υπάρχουν, ε, ξέρετε, και κάποιες ε, φιλικές διαδικασίες στη Γαλλία, συνενετικές, που δεν περιλαμβάνονται βέβαια σε αυτή την πρόταση οδηγίας, όμως στη Γαλλία έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικές για την εξέβρεση λύσεων αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα με νούμερα κιόλα. Ε, οι διαδικασίες αυτές ε, οι φιλικές προβλέπουν γρήγορο διακανονισμό ε, για έξοδο των επιχειρήσεων από την κρίση. Το 2016 είχαμε γύρω στις 2.500 τέτοιες διαδικασίες που έσωσαν 612.000 θέσεις εργασίας. Αν το συγκρίνουμε με τις δικαστικές εκαθαρίες που είχαμε στη Γαλλία 43.000 ε, τον αριθμό. Αυτές αφορούσαν 107.000 θέσεις εργασίας που ακριβώς δυστυχώς επειδή υπήρχε πάυση δραστηριότητας και καθάριση χάθηκαν. Απελήθησαν οι εργαζόμενοι αυτοί. Και βλέπετε ότι η επιτυχία αυτών των φιλικών δικανοσμών είναι κάτι πολύ θετικό, γιατί διατηρούνται θέσεις εργασίας και παραμένουν οι επιχειρήσεις. Ε, στην οικονομία και καταλάβαμε ότι μπορεί αυτό να περιλαμβάνεται στην πρόταση της οδηγίας, όμως ε, αυτά τα σχήματα, αυτά τα προγράμματα που προτείνουν θα μπορούσαν να συνδεθούν με την παράλληλη ύπαρξη. Δηλαδή να έχουμε και αυτά στους ε, φιλικούς διακανονισμούς και αυτά που προβλέπει η οδηγία ως διαδικασίες. Είμαστε επίσης ε, υπέρ και σύμφωνα με το γεγονός ε, ο φιλέτης ε, να μην, να μην του παίρνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Υπάρχει η, η επιταχυμένη διαδικασία διάσωσης και η διαδικασία διάσωση απλή. Όταν συμφωνήσουν περισσότεροι πιστωτές μπορεί να υπάρξει ουσιαστικά μία μη λήψη υπόψη των λιγότερο σημαντικών πιστωτών, κάτι που λέγεται cross-class cram-down. Αυτό δεν μας βρίσκει βέβαια σύμφωνος. Ε, συμφωνούμε τώρα με τον δεύτερο άξονα για να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στα φυσικά πρόσωπα, έτοιμους επιχειρηματίες. Εμείς έχουμε δύο λύσεις στο γαλλικό σύστημα, σε αυτή την πρόταση. Πρώτα απ' όλα, οι δικαστικέ εκαθαρίσει οδηγούν σε καθάριση και του χρέου. Και στην τελευταία μεταρρύθμιση που κάναμε, ε, υπήρξε επιτάχυση των διαδικασιών με τις δικαστικές απλουστευμένες εκαθαρίσει, ε, με την προθεσμία να είναι λιγότερο από δύο χρόνια για την επεξεργασία. Σε ό,τι δε αφορά το διάταγμα του 12 Μαρτίου του 2014, η διαμερομηνιακή σύσταση. Εδώ δημιουργούμε τη διαδικασία από αποκατάστασης ώστε ένα φυσικό πρόσωπο με ενεργητικό κάτω των 5.000 να μπορεί να, να απολαμβάνει κατάργηση του χρέους του μέσα σε πέντε μήνες. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μέτρα για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συλλογικών διαδικασιών, νομίζω ότι εμείς συμφωνούμε με τις διατάξεις του, έχουμε τον νόμο Μακρόν, για την εξειδίκευση, την κατάρτιση των δικαστών, δημιουργούνται εξειδικευμένα εμποροδικεία. Επίσης έχουμε το νόμο εξυγχρονισμού της δικαιοσύνης 18 Νοεμβρίου του 2016, 21 για την επιτάχυνση της κατάρτισης κάποιων άλλων ε, δικαστών. Δημιουργείται και μια ηλεκτρονική πύλη για την ε, διαβίβαση όλων αυτών των στοιχείων, όπως είναι οι απαιτήσει των ε, πιστωτών, κοινοποίηση του σοφλέτς κτλ. κτλ. Θα γίνουν κάποιες προσαρμογές, αλλά νομίζω ότι θα είναι εύκολες. Και τέλος, ότι αυτά τα στατιστικά δεδομένα, το, Εθνικό, το Συμβούλιο Επικρατείας το Εθνικό Μάλλον Συμβούλιο έχει κάποια στοιχεία τα οποία όλοι μπορούν, στα οποία όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση. Έχω δύο λεπτά για να σα μιλήσω για τι απαιτούμενε προσαρμογέ. Εμεί θεωρούμε ότι το πεδίο εφαρμογή για τα άρθρα 1 και 4 χρήζει περαιτέρω διευκρινήσεων συγκεκριμένα. Το πενδεχόμενο αφαιρεγγιότητας ε, νομίζω ότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ε, δυνατοτήτων και πιθανοτήτων. Θα πρέπει να δούμε ίσως ε, πάλι ε, το, το θέμα των ε, συνδίκων και τα λοιπά και τα είπε και ο προλαλής σας, αν μπορεί ο ίδιος ο επικαιρμητής να ορίζει για όλες τις διαδικασίες. Επίσης έχουμε ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά το βολονταριστικό χαρακτήρα της διαδικασίας. Δηλαδή, στο δικό μας σύστημα, ε, ο φιλέτης είναι αυτός ο οποίος ζητά ε, την προστασία του δικαστηρίου και αυτό γίνεται σε πρόωρο στάδιο. Δηλαδή, από τον ίδιο κινείται η όλη διαδικασία. Το να μπορούν να το κάνουν αυτό και οι πιστωτές μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Τέλο, η μείωση της μέγιστης διάρκεια περίοδου παρατήρησης 18 σε 12 μήνε και αυτό μα δημιουργεί ένα πρόβλημα με τι διαδικασίε διάσωση, γιατί η περίοδο παρατήρηση για μα ανέρχεται σε 18 μήνες και όχι 12, αλλά και εδώ μπορούμε να το δούμε και να εξελιχθούμε και εμείς ίσως. Ε, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης βέβαια, χάρη στην οδηγία γενικά και επίσης θεωρούμε ότι για να υπάρξει αναρμόνιση με το γαλλικό δίκαιο ε, μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές με ευέλικτο τρόπο και να καταλήξουμε σε ένα απόλυτα εναρμονισμένο σύστημα, ε, εναρμονισμένο με τους στόχους της οδηγίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστούμε. Έχουμε τώρα κάποιο χρόνο για συζήτηση. Υπάρχουν τίποτε ερωτήσεις που θέλετε να θέσετε, κυρία Ρέγνερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ε, παρουσιάσεις. Δείχνει το πόσο προσεκτικές ρυθμίσεις απαιτούνται αν θέλουμε να έχουμε αυτό το καστός της δεύτερης ευκαιρίας. Το ερώτημά μου απευθύνεται πρώτα απ' όλα στον κύριο Μπίρμπαχ. Αναφέρατε συγκεκριμένες πτυχές που δεν γνώριζα Δηλαδή για εμένα πάντα το θέμα ήταν να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τους ασθενέστερους αυτούς που χρειαζόταν προστασία. Αυτό πρέπει να είναι πάντα αυτό το οποίο λέμε. Αλλά εσείς αναφερθήκατε στην σταθερότητα των χρηματαγορών ε, και την πτυχή στη γενικότερη, τη ματιά στη γενικότερη οικονομία. Γι' αυτό το ερώτημά μου αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία αναφέρατε. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, πλήττονται περισσότερο από άλλες, υπάρχουν κλάδοι που πλήττονται περισσότερο από άλλους ή είναι μεικτή εικόνα. Γιατί αυτό το οποίο αναφέρατε είναι πάρα πολύ συναρπαστικό. Ότι δηλαδή πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ Και βεβαίω τώρα υπάρχουν οι λομπίστες για τις ε, τράπεζες, αλλά βλέπουμε πως οι τράπεζες, ειδικά οι μικρές τράπεζες, γνωρίζουν καλύτερα ε, τους ε, πελάτες τους ε, και γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν στην περίπτωση αναδιάρθρωσης. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη για το αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τι γίνεται με τα ταβάνια αυτά πολλούνται σε άλλους, ποια είναι η γενική εικόνα θα λέγατε, για την σταθερότητα του κλάδου αυτού. Νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο ολόκληρης της ε, εσωτερικής αγοράς. Ε, δηλαδή ακούγεται κάτι πάρα πολύ ωραίο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Σας ευχαριστώ κυρία Νίμπλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω ε, τους ε, συναδέλφους που έκαναν εδώ πέρα τις παρουσιάσεις. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να τους ευχαριστήσω. Τώρα δεν θα, δεν ε, θα σχολιάσω. Έχω την δυνατότητα στο τέλος ως συγκήτρια να μιλήσω πέντε λεπτά. Έχω λοιπόν δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτη μου ερώτηση. Με ενδιαφέρει να μάθω. Θεωρείτε πως η πρόταση έχει ρυθμιστεί αρκετά για το πώς, πότε μπορούν να ξεκινήσουν διαδικασίες αναδιάρθρωση. Ε, με ότι όταν ε, ένας οφειλέτης έχει οικονομικές ε, δυσκολίες ε, θα πρέπει να μπορεί να επιλέγει, λέτε, πρώτο ερώτημα. Δεύτερον, άκουσα ότι 80% των χροκοπιών οφείλονται σε αποτυχίες της διοίκησης. 80% για τον οποιονδήποτε λόγο. Εάν λοιπόν ισχύει κάτι τέτοιο, έχει νόημα οι πιστωτές ε, και οι οφειλέτες να φτάσουν σε αυτή τη διαδικασία. Μήπως θα έπρεπε πολύ νωρίτερα στην διαδικασία αυτή να εμπλακεί κάποιος ειδικό είτε τον ορίσει το δικαστήριο είτε όχι, είτε είναι ένας ε, ειδικευμένο σε αυτά τα ζητήματα, ένας ουδέτερος τρίτος αντικειμενικός, σε πάση περιπτώσει, να προσπαθήσει να βρει την σωστή ισορροπία μεταξύ των ε, διαφορετικών συμφερόντων. Θα ήθελα να ακούσω και την άποψή σας από αυτού. Τρίτη ερώτηση. Έχω πολλές ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Τα περιοριστώ σε αυτές. Ε, cross-class cram down. Άκουσα πάρα πολλά πράγματα και κριτική κυρίως γι' αυτό. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να ληφθεί μία απόφαση για ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης. Ε, αν γίνει η διαδικασία όπως προβλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, αν δεν σας αρέσει αυτή η διαδικασία, ποιες είναι οι δικές σας οι προτάσεις ή θα πρέπει απλά να περιμένουμε τις αποφάσεις ανακατηγορία πιστωτών ε, για να φτάσουμε στο τέλος. Ε, θα ήθελα να ακούσω την δική σας την πρόταση. Και αν έχουμε χρόνο να ξανακάνω ερωτήσεις. Αλλά φαντάζομαι θέλει να μιλήσει για κάποιος άλλος. Thank you as well. Ε, Mrs. Lopez Bermego. Η κυρία Λόπεθ Μπερμέχο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους προσκεκλημένους για τις εισηγήσεις τους που ήταν πολύ συγκεκριμένες και διαφώτισαν πολλές πτυχές του θέματος. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω στην άποψη της ΕΤΟΚ που λέει ε, τι ανησυχεί για την πρόταση της οδηγίας σε περί αφαιρεγκαιότητα που αγνοεί συγγνώμη, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Εγώ νομίζω ότι αυτό που απαιτείται είναι ένας καλύτερος ορισμός, ώστε οι επιχειρηματίες και οι τράπεζε να μην συμφωνούν ε, για αποπληρωμή των χρεών ε, και για εκπλήρωση των απαιτήσεών του σε βάρος ακριβώς των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν θέλω να επιμείνω. Υπάρχουν ε, τροπολογίε και από την Επιτροπή Εργασία και από την Επιτροπή συγγνώμη, και την Επιτροπή των Οικονομικών. Σε τι τακτικέ πτωχεύσει, έχω ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα και μπορείτε να απαντήσετε στη συνέχεια. Θεωρείτε δηλαδή ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το κείμενο για να αποφευχθεί το γεγονό αδίστακτε επιχειρήσει να χειραγωγούν τα στοιχεία του, οικονομικού λογαριασμού του, ε, ώστε τα έσοδά του ε, να τα πηγαίνουν ε, σε θηγατρικέ για να δικαιολογήσουν μαζικέ απολύσει ή μονομερή αλλαγή των εργασιακών συνθηκών αν δεν αλλάξουν βέβαια οι αντικειμενικές συνθήκες παραγωγής. Εγώ γνωρίζω δυστυχώς ότι υπήρξαν τέτοιε περιπτώσεις και θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς και εσεί τι πιστεύετε. Η κυρία Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις αυτές, οι οποίες όλες μου φάνηκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, αλλά πραγματικά ε, εγώ και από την ε, δική μου σταδιοδρομία, 35 χρόνια απασχολήθηκα με την αφαιρεγκαιότητα και μετά από 35 χρόνια δουλειά στην δικασία αφαιρεγκαιότητα της δική μου περίπτωση, το πρόβλημά μου δεν ήταν μόνο η τραπεζική εγγύηση, αλλά και το leasing. Οι μικρές εταιρείες αυτή τη στιγμή, ιδίως οι γεωργικές εταιρείες, οδηγούνται σε αφαιρεγγιότητα διότι τα υλικά περιουσιακά του στοιχεία ε, ανήκουν σε μια τράπεζα με, την, ε, με το leasing, την εκμίσθωση. Από τη στιγμή που υπάρχει πάυση πληρωμών, ε, δηλαδή δεν μπορούν να πληρώσουν το νίκη τους ή τα δανειά τους οι εταιρείε και πρέπει να παραδώσουν και να ξεκινήσουν τη διαδικασία της αφαιρεγγιότητας με την προστασία κάποιου δανειστή, ε, τότε η εταιρεία του leasing, δηλαδή η τράπεζα, ξαναπαίρνει πίσω τα υλικά περιουσιακά στοιχεία και τα πουλάει για δικό της λογαριασμό, παίρνοντας ταυτόχρονα και τα νίκια του ανθρώπου αυτού που αναγκάζεται να ε, δηλώσει πτώχευση. Το βρίσκω καθαρή απάτη, διότι η τράπεζα από τη μια και, πληρώ, και πουλάει τα υλικά αγαθά και τα ξαναγοράζει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα του leasing, της εκμίστοσης. Θα πρέπει να το δούμε με πολύ αυστηρό τρόπο, να μην μπορεί δηλαδή κανείς να αγοράσει υλικά ε, αγαθά που τα αγοράζει κανείς το 60-80% της ε, τιμής. Ε, εδώ η εταιρεία δεν μπορεί να ξαναστεθεί στα πόδια της προφανώς μετά από αυτό. Πού είναι η δεύτερη ευκαιρία για την οποία συζητάμε και το άλλο που πάντοτε με ανησυχούσε ήταν ότι οι τράπεζες δανείζουν τις εταιρείε, βεβαίως, εταιρείε που είναι, έχουν αυτό το νομικό καθεστώς αλλά ζητώντα την προσωπική εγγύηση του διαχειριστού. Αυτό σημαίνει ότι η πτώχευση μπορεί να περάσει και μετά ε, υπάρχει η δίωξη κατά του ίδιου του εγγυητή. Πού θα έφερε τη δεύτερη ευκαιρία αυτό ο Γιώργο που θα του πουλήσουν τα υλικά περιουσιακά του στοιχεία, τα έχει παρελάει η τράπεζα και μπορεί να προσπαθήσει να ξαναρχίσει την οικονομική του δραστηριότητα, αλλά διώκεται νομικά για την δική του αφαιρεγκαιότητα πλέον από την τράπεζα. Δεν θέλω να ε, γίνω ιδεαλίστρια, αλλά η πραγματικότητα των ε, πτωχεύσεων είναι αυτή. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου. Οι αξιότιμοι προσκεκλημένοι μας θα επιθυμούσαν να απαντήσουν ποιος θα ξεκινήσει. Επειδή μου ετέθη ένα συγκεκριμένο ερώτημα, θα ξεκινήσω εγώ σε ό,τι αφορά αυτέ τι πτωχεύσει για λόγου τακτική. Ε, και τι, πώς μπορούν να αντιδράσουν οι εργαζόμενοι, εκπρόσωποι των εργαζομένων ε, συγκεκριμένα, Μπορώ να δώσω μια πολύ σαφή απάντηση, διότι το συνδικαλιστικό κίνημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει εξεργαστεί το θέμα και έχει συζητήσει ευρέως ε, το τι πρέπει να γίνει και είναι η πρώτη φορά που υπήρξε μια απόφαση ε, που λέμε πλέον ότι σε όλες τις επιχειρήσεις από 200 και πάνω μισθωτούς κάποιοι ξεκινούσαν και από τους 50 τέλος πάντων και μπορεί και από τους 50 να υπάρχει εκπροσώπηση των εργαζομένων αυτή είναι η διαπραγματευτική μας θέση αλλά λέμε ότι στις μικρές επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να επηρεάζουν τα πράγματα και τα πράγματα βέβαια στην Ευρώπη διαφορετικά. Υπάρχει πάντως αυτή η εκπροσώπηση και εμείς θέλουμε μία μόνιμη εκπροσώπηση των, ε, των εργαζομένων σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα, να υπάρχει δηλαδή το μόνιμο δικαίωμα διαβούλευσης και ενημέρωσης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αποτρέψουμε εμείς το ενδεχόμενο τέτοιων πτωχεύσεων για λόγους τακτικής ε, και οι εγκληματίες, ε, όποιοι, πώς και οποιονδήποτε άλλο νόμο, έτσι και αυτό το νόμο μπορούν να τον παραβιάσουν αν θέλουν. Αλλά σε ό,τι αφορά την πρόσβαση, αυτή είναι πιο εντατική και υπάρχουν δυνατότητες επιρροής ε, των αποφάσεων από τους τα εργασιακά συμβούλια, τι επιτροπέ επιχείρηση, από του εργαζομένου, εκπροσώπου του. Ε, αυτό είναι κάτι που δεν έχει προηγούμενο ε, και αυτό που ζητούμε είναι η μόνιμη εκπροσώπηση και μάλλον συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στι οικονομικέ διαδικασίε. Ένα είδο ε, δηλαδή οικονομική επιτροπή που θέλουμε να καθιδρυθεί στα επιχειρήσει για την κυρία Νίπλερ που είπε πότε μπορεί να ξεκινήσουν. Αν το συνδέσω με τους ε, συνδικαλιστές και τους εκπροσώπους των εργαζομένων, όπου θέλουμε να έχουν ε, και αυτοί το λόγο στη ε, εξαγωγή των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης και αν δούμε και τη σχέση της ε, διοίκησης με τους ε, εκπροσώπους των εργαζομένων για την επίτευξη συνένεσης. Ναι, ε, να συμφωνήσουμε πότε είναι ανάγκη να ξεκινήσει η διαδικασία αναδιάρθρωσης, να κατατεθεί έτοιμα κτλ. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της διοίκησης και αυτό να ε, αποτελεί το έναυσμα για να ξεκινήσει η διαδικασία της αναδιάρθρωσης, για να τις στην για την έναρξη. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει και τώρα για ουδέτερες αντικειμενικές, ε, αδικές, ουδέτερες αντικειμενικούς φορείς. Ναι, πράγματι ε, είναι πρόδειλο ποιοι μπορεί να είναι αυτοί οι μεμονωμένοι φορείς. Αν υπάρχει αναγκαιότητα, νομίζω ότι ναι μπορεί να γίνει και έτσι και εμείς βλέπουμε τα πράγματα. Για το τελευταίο, κυρία Λελού Τομά, συμφωνούμε απόλυτα με τον διορισμό ενός ανεξάρτητου οργάνου που θα αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα. Είναι απολύτως αναγκαίο κάτι τέτοιο. Τα κράτη πρέπει να αποφασίζουν αν θα είναι διοικητικό ή δικαστικό ο φορέα αυτό, αλλά είναι κατά μα πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί αυτό το όργανο. Σε ό,τι αφορά το leasing, ε, αν με πρέπει να δώσω το λόγο στην ωραία Περντερό, τη συνάδελφό μου για να μιλήσει για τα σχετικά με τους δημοκράτες. Ε, Ευχαριστώ. Μια τεχνική διευκρίνηση για την ε, τύχη των υλικών περιουσιακών στοιχείων στην περίπτωση του leasing. Το πλαίσιο προβλέπεται από την οδηγία και προβλέπεται και από τους κανόνες για την ε, προστασία της γαλλικής νομοθεσίας Εάν φαίνεται βιώσιμη διαδικασία, ο εκαθαριστής μπορεί να εξαναγκάσει στην πώληση των περιουσιακών στοιχείων το άλλο μέρος της ε, σύμβασης εκμίσθωσης, κάτι που μπορεί να συμβεί αν υπάρχουν απλήρωτα ποσά πριν την έναρξη της διαδικασίας αφαιρεγγιότητας, δηλαδή να απαιτήσει την εκτέλεση των συμβασιακών υποχρεώσεων, δηλαδή να αποπληρώσει λόγου χάρη τα ενίκια, πληρών, πολλώντας τα υλικά περιουσιακά στοιχεία. Στην περίπτωση λοιπόν που η δραστηριότητα έχει πάυσει, είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εφόσον η δραστηριότητα συνεχίζεται, τα συμβόλαια μπορούν να συνεχίσουν να ισχύουν και να απαιτείται η εκτέλεσή τους. Μια πληρωματική παρατήρηση για το θέμα των κριτηρίων για να οριστεί το σημείο αφετηρίας ε, και έναρξης της διαδικασία ε, αναδιάρθρωσης. Είναι σημαντικό να δούμε ότι υπάρχουν διαφορετικέ περιπτώσεις εδώ ανάλογα με το εάν ο δανειστή ε, θα ζητήσει να υπάρξει δίωξη ή όχι. Εάν η αναστολή αυτών. Εάν υπάρξει αναστολή της δίωξης, εδώ μιλάμε για σοβαρές δυσκολίες που δεν μπορούν να, να τις ξεπεράσει η εταιρεία. Δυσκολίες που απουσία της αναστολής δίωξης μακροπρόθεσμα απομακρύνει πολύ από την κατάσταση της αφαιρεγγιότητας. Ευχαριστώ από τη ΓΟΑΠΜΕ. Παρόλο που δεν έγινε συγκεκριμένη ερώτηση προς εμένα, θέλω να πω τη γνώμη μου. Τις τεχνικές διευκρινήσεις για την αφαιρεγγιότητα. Η πρόταση αυτή νομίζω πετυχαίνει πολύ σωστό σημείο ισορροπία όταν προσπαθεί να συμφιλειώσει τις διαφορετικές εθνικές νομοθεσίε Και αν θέλουμε να πάμε μακρύτερα σε εθνικό επίπεδο, πρέπει να προβλέψουμε μέτρα για να διευθετήσουμε και τεχνικώ την, την αφαιρεγκαιότητα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω ότι υπήρχε κάποια συμφωνία για τα βασικά σημεία και επιπροσθέτως δεν είναι οδηγία ακριβώς εναρμόνισης λόγου χάρη η κατάταξη των αξιολογήσεων είναι δυνατόν να βρεθεί εδώ ευρωπαϊκή λύση, να υπάρξει απόλυτη συμφωνία για το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε δεν το λύνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά τα άλλα, δεν κατάλαβα πολύ καλά αυτό που είπε ο συνάδελφο από τις συνδικαλιστικέ οργανώσεις. Γιατί μιλούσατε στα αυτή μου και προσπαθούσα να ακούσω τη διερμηνία. Δεν είναι εδώ το μέρος για να προβλέψουμε νέους κανόνες για την εκπροσώπηση των εργαζομένων. Εάν διαβάσετε προσεκτικά την πρόταση, υπάρχουν πολλές αναφορές, πολλές εγγύησεις ήδη, αν και ίσως εγώ σας παρανόησα, οπότε να με συμπαθάτε, και πραγματικά απευθύνω έκκληση προς το Ευρωκοινοβούλιο να ακολουθήσει μια ήπια προσέγγιση. Σκεφτείτε την πλειονότητα των επιχειρήσεων που είναι μικρό και με, ε, επιχειρήσεις και τι θέλετε να πετύχετε αναφερόντως αυτή την οδηγία. Δεν πρέπει να δυσχεράνουμε περαιτέρω τις διάφορες διαδικασίες, διότι ούτως ή άλλως πολλές φορές και χρονοβόρες είναι και δαπανηρές για τις εταιρείε. Και καλό είναι να σκεφτόμαστε πρώτα τους μικρούς στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ich will versuchen, kurz auf alle Fragen einzugehen, bei denen ich mich angesprochen fühle. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Μια ερώτηση ήταν αν θα φοβόμαστε ότι θα αυξηθούν τα μη εξπερτούμενα δάνεια. Η πρόταση εδώ ουσιαστικά έχει να κάνει με την ανάγκη να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες. Ε, μετά από τη χρηματοπιστωτική κρίση ε, υπήρξε αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία ε, όλο και περισσότερο αυξάνονται, σωρεύονται και η αφαιριότητα και οι διαδικασίες δεν, λειτουργεί καλά, το, δεν λειτουργούν καλά, γι' αυτό και χάνονται πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Γι' αυτό εμείς λέμε να περιορίζεται αυτό το, αυτή η οδηγία μόνο στους πιστωτές στον τομέα το πιστωτικό, σε ό,τι αφορά τις μικρότερες ε, τράπεζες που χρηματοδοτούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ε, είναι κάτι σημαντικό. Μια τράπεζα έχει ε, τελείως διαφορετικά ενδιαφέροντα και βλέπει τελείως διαφορετικά αν είναι επιτόπου ε, τον ε, εργαζόμενο από μια μεγάλη εμπορική τράπεζα που έχει την έδρα της στο Λονδίνο ή στη Φραγκφούρτη και τελείως διαφορετικά κριτήρια για τη χρηματοδότηση. Αυτά δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε, ότι εμείς αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι ένα εργαλείο ώστε να βοηθηθεί η χρηματοδότηση αυτών των μικρών επιχειρήσεων. Για το πότε πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία ε, αναδιάθεσης που είπε η κυρία Νίβλε. Νομίζω ότι υπάρχει πρόταση. Ε, αν δεν υπάρχει λόγος, δεν μπορεί να κινηθεί αυτή η διαδικασία. θα πρέπει να τηρηθούν οι ε, εθνικές αλλά και οι ευρωπαϊκές διαταξένα. Ένα εσωτερικό όριο πρέπει να υπάρχει. Ας πούμε ότι αύριο εγώ πτωχεύω, έχω τέσσερις μήνες μορατόριο, το οποίο μπορεί μετά να επικοινωνηθεί. Δεν μπορούν ε, παρά και τα δύο να λαμβάνονται υπόψη. Πρέπει να υπάρχει το εσωτερικό όριο κατά την άποψή μου. Σε αυτό ε, το ποσοστό, το 80% που λέτε ότι εκεί έχει αποτύχει τελικά η διοίκηση, ναι, πράγματι αν δεν υπάρχει ένας ουδέτερο ε, φορέας επίσης δεν μπορεί, να δεν μπορεί να διορθωθεί το πρόβλημα γιατί χρειάζεται επιτήρηση, χρειάζεται και ενίσχυση, στήριξη. Είναι τελείως ε, ίδια τα πράγματα σε Γερμανία και Γαλλία. Αν ένα σύνδικο λέει το κοίταξα, μπορείς ε, να συνεχίσεις, έχεις μια δεύτερη ευκαιρία, μπορείς να επιβιώσει. Αυτό είναι τελείω διαφορετικό από το αν δεν υπάρχει καμία υποστήριξη. Όλοι οι συμμετέχοντες και οι πιστωτέ χρειάζονται διαφάνεια και πολλές φορές δεν λαμβάνουν λογικέ αποφάσει ή επιχειρήσει όταν τίθεται θέμα ζωή ή θανάτου για αυτές. Αυτό είναι γεγονό. Για το leasing ε, και τις εγγύσει για τι επιχειρήσει, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό στην πρόταση τη Κομισιόν. Μιλάμε για την ε, πτώχεια μιας επιχείρησης ή την υπεραίωση μιας επιχείρησης. Τι γίνεται όμως με την εγγύηση. Δεν ε, το ε, επηρεάζει αυτό η συγκεκριμένη πρόταση. Δεν το θίγει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε και αυτά τα θέματα των εγγύησεων. Ευχαριστώ κυρία Γκάιο. Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Τρία λεπτά, δεν έχετε παραπάνω. Σύντομα. Θα απαντήσω στα ισπανικά στις γενικές ερωτήσεις και στη συγκεκριμένη ερώτηση της εισηγήτριας σε άλλη γλώσσα. Λοιπόν, πότε να ξεκινούν οι αναδιαρθρώσεις της κυρίας Νίμπλερ ερώτηση. Εγώ με το λάκη Χουντόβιν δεν έχω πρόβλημα, σας πω την αλήθεια, γιατί ούτως ή άλλως θα πρέπει ε, να ληφθούν οι αποφάσεις και χρηματοπιστωτικοί φορείς. Ε, θα είμαστε οι πρώτοι που θα αναλύσουμε την κατάσταση, θα κάνουμε τη μελέτη του ολογισμού της επιχείρησης και θα δούμε κατά πόσον ε, χρειάζεται να γίνει μια θυσία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Άρα το likelihood, η πιθανότητα, νομίζω ότι είναι λογικό ως κριτήριο, ό,τι αφορά το ποσοστό το 80% της ευθύνης της διοίκησης. Δεν ήξερα εγώ αυτό το ποσοστό. Και αυτό έχει να κάνει και με αυτά που απάντησαν ε, οι συνάδελφοι από τη Γαλλία και τη Γερμανία, που είναι σύνδικοι. Ε, αυτό που έχω να πω για την Ισπανία, το είπα και στην αρχή, εμείς έχουμε ένα ιδιωτικό μοντέλο, ε, αμυγός ιδιωτικό. Δεν παρεμβαίνει κανένας ε, διαχειριστής, κανένας από τη διοίκηση και λειτουργεί αυτό το μοντέλο. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι καλό το γαλλικό, το γερμανικό μοντέλο και σίγουρα είναι πάρα πολύ καλά αυτά τα μοντέλα. Εγώ απλά θέλω να τονίσω ότι όλα αυτά έχουν ένα κόστος και σε κάποιες περιπτώσεις το κόστος αυτό ίσως να μην μπορεί κάποιος να το επομιστεί. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιβάλλουμε αυτό το μοντέλο, αυτό πρέπει να το δούμε. Η ισπανική μου εμπειρία μου λέει ότι μέχρι τώρα είναι πολύ επιτυχημένο το δικό μας μοντέλο. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις για το cross-class cram-down, το είπα και στην παρέμβασή μου στην ε, Ισπανία, δεν το έχουμε το cross-class. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι ότι είμαστε και κάθετα αντίθετοι, ε, αυτό μπορούμε να το δεχθούμε. Το cram up μας ανησυχεί όμως, αυτό που το είπα, δηλαδή να χάσουμε την ασφάλεια δικαίου σε ό,τι αφορά ε, την κατηγοριοποίηση των πιστωτών. Αυτό να μην το ορίζουν οι νόμοι, αλλά οι πιστωτές. Αυτό σημαίνει μείωση της ασφάλειας δικαίου και θα επηρεάσει και την τιμή. Άμεσα θα επηρεάσει την τιμή των πιστώσεων. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση της σα της κυρίας Λόπεθ Μπερμέχο για τα δικαιώματα των εργαζομένων, απάντησαν ορισμένοι από τους απελαρίσαντες ε, συναδέλφους. Ακούστε, μας είπε η κυρία Λόπεθ Μπερμέχο ότι ξέρει τέτοιες ε, περιπτώσεις ε, ε, που ήταν δόλια ε, και για λόγους τακτικής η πτώχευση. Εγώ δεν τα ξέρω, δεν έχω συμμετάσχει σε κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής. Θέλω να σας πω επίσης, και το ξέρετε φαντάζομαι, ότι το 2015 ορίστηκε η ποινική ευθύνη νομικού προσώπου. Όχι μόνο διαχείριση της τράπεζας που αρεμβαίνει στις επιχειρήσεις ε, αυτές, αλλά και του νομικού προσώπου. Αν υπήρχαν λοιπόν ήδη κάποιες εγγύησεις και κάποιες προφυλάξεις, ακριβώς για να τα αποφύγουμε αυτά γιατί στη δική μου τη ένωση εγώ είμαι υπέρ. Για να έχουμε λοιπόν τέτοιες ε, τα, τακτικές τώρα έχουν ενισχυθεί αυτές οι, αυτά τα ηχέγγυα και επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω ότι φυσικά και πιστεύω ότι όλοι οι stakeholders όπως τους λέμε ανησυχούν και ενδιαφέρονται για τον εργαζόμενο και η τράπεζα. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι να μην μπορούν να το αντιληφθούν αυτό, να δυσκολεύονται να το καταλάβουν, αλλά είμαστε όλοι ε, ε, έχουμε επίκεντρο τον εργαζόμενο και στην περίπτωση πτωχεύσεων, εκαθαρίσεων. Ένα θέμα, δεν ξέρω, απάντησα την ερώτησή σας ή όχι. Ίσως κάτι δεν κατάλαβα καλά. Ε, ε για αν υπάρχει, το αν υπάρχουν κίνδυνο για περισσότερα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όχι, γιατί πότε έχουμε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όταν πτωχεύουν οι επιχειρήσει. Αν εμεί μπορούμε να κάνουμε μια θυσία και να σώσουμε του πελάτε μα στην προκειμένη περίπτωση, τότε νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των μη εξυπηρετούμενων αν έχουμε αντιδράσει και Thank you very much. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος χρόνος Μια άλλα σχόλια. Η κυρία Νίμπλερ τώρα θα κάνει τις τελικές της παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια που έχει προχωρήσει η ώρα, θα περιοριστώ σε 4-5 παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τους ε, ειδικού μας. Δεύτερον, Και λαμβάνω υπόψη ότι ο κύριο Χέντριξ ε, έθεσε τα πράγματα διαφορετικά από τον κύριο Μπίμπαχ όσον αφορά το φάσμα. Τρίτον, για εμένα νομίζω είναι σημαντικό να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων πιστωτών οφειλετών εργαζομένων. Πρέπει να δούμε πώς θα βρεθεί η ισορροπία αυτή, μήπως είναι πολύ φιλικοί στους οφειλέτες, πολύ φιλικοί στους πιστωτές, είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Τέταρτον, γνωρίζω, υπάρχουν και κίνδυνοι και ευκαιρίες και δυνατότητες περαιτέρω οικονομικής επιτυχίας αλλά και κίνδυνοι όπως είπαμε θέμα, αναφέρθηκε το θέμα των τακτικών χρεοκοπιών ή δευτερογενών χρεοκοπιών των προμηθευτών μιας επιχείρησης. Ακούστηκαν πάρα πολλά για την έννοια του λεγόμενου τίμιου επιχειρηματία αυτό το οποίο εσείς αναφέρατε πράγματι πάρα πολύ σημαντικό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, τελευταίο διάβολος ε, κρύβεται στις λεπτομέρειες. έχετε ε, δίκιο, εσείς έχετε μια διαφορετική διαδικασία. Επίση θέλετε να γίνουν πιο συγκεκριμένα τα πράγματα, ειδικά όσον αφορά τις προθεσμίες ε, και την απαλλαγή. Το θέμα του cram down επίσης πρέπει να το δούμε. Και πολλές άλλες ε, λεπτομέρειες. να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποια ισορροπία. Θα πάμε λοιπόν νομίζω στις ε, διαβουλεύσεις. Και να δούμε το τι θα πάει μετά στην... πριν πάντα πράγματα στην μετάφραση τα κείμενα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much for this closing... Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις καταληκτήριες ε, παρατηρήσεις σας. Να ευχαριστήσω τους αξιότιμους μας, προσκεκλημένους μας σήμερα να ε, κλείσουμε αυτή τη συνεδρίαση και να θυμίσω στους συναδέλφους ότι στις 4.30 έχουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ε, ακρόαση για τις δυνατότητες και προκλήσεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο σημερινό μεταναστευτικό πλαίσιο. Είμαι ε, απολύτως βέβαιος ότι θα είστε όλοι εδώ για αυτή την ε, ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ.